Good morning everyone. Καλημέρα σας. Η μερίσια διάταξη μερικής μας συνεδρίασης την έχετε λάβει. No, this is afterwards. But you, we have to approve the agenda. Okay, so you received the agenda of today. Έχετε λάβει τη σημερινή συνεδρίαση, τη μερίσια διάταξη. Ανακοινώσεις προτείνω να κάνουμε μετά τις ψηφοφορίες που έχουμε λιγότερη χρονική πίεση. Πρακτικά έχετε 20-21 Ιουνίου. Αν δεν κατατεθούν σχόλια μέχρι το τέλος της ε, σημερινής μας ημέρας και συνεδρίασης εγκρίνονται. έκθεση ε, πεπραγμένου σε σχέση με τις αναξελίξει διοργανικές ε, διαπραγματεύσεις. Πάλι θα τη δούμε μετά τις ψηφοφορίες και έτσι πάμε στο FG72 ε, κάθετος 4406 ε, γενετικά τροποποιημένη φασίου λισόγιας για να δούμε να μας πει ο κύριος Φρόντε, νομίζω ότι σαν τον κύριο Πρόντσε. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Όπως είπατε, εκπροσωπώ τον Μπάρτ Στάις, που είναι στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Σας διαβάζω ένα κείμενο το οποίο έχει ο ίδιος ετοιμάσει όμως. Λοιπόν, σήμερα συζητούμε αυτά τα δύο σημεία των αντιρρήσεων για τους γενετικά τροποποιημένους σπόρους υφασιορούς σόγιας που έχουν υποστηρίξει και διάφορες ε, άλλε επιτροπέ. Έχει δώσει μια θετική γνώμη, εκδώσει μια θετική γνώμη η ΕΦΣΑ, αλλά τα κράτη-μέλη έχουν προβάλει αντιρρήσεις λέγοντας ότι για το φαινοτυπικό, φαινοτυπικά στοιχεία δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες, ε, τοξικολογικά στοιχεία δεν είναι επαρκή, γιατί το υποχρονία τοξικότητα έχουμε μια δοκιμή μόνο 70 ημερών που δεν αρκεί και είναι πολλά τα κράτη-μέλη που ανησυχούν για την ε, απόφαση αυτή της ΕΦΣΑ. Αποτελέσματα της μόνιμης επιτροπής ε, και της Επιτροπής Προσφυγών για, τις, ε, για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς δεν έχουν ληφθεί υπόψη, δεν έχει εξασφαλιστεί ειδική πλειοψηφία για να περάσει αυτή η υπόθεση από τη μόνιμη επιτροπή. Μόνο 10 κράτη-μέλη την υποστήριξαν και η αξιολόγηση του κινδύνου από πλευρά ΕΦΣΑ δεν αρκεί όπως μας λένε τα κράτη-μέλη γιατί δεν ε, ικανοποιούνται με λύματα σχετικά με ε, κρεμότητες, αβεβαιότητες και συνέπειες στο ανοσοποιητικό και το ε, αναπαραγωγικό σύστημα. Στην γλυφοζάτη, τη γλυφασινάτη, γλυφοζάτη, γλυφοζινάτη ή και άλλες ουσίες, ε, συνολικά τρία είναι τα, οι κυρίες ομάδες προϊόντων στις οποίες εμφανίζονται, σε ζυζανιοκτώνα δηλαδή, ε, με συνέπεια να ανοιχνεύονται στη συνέχεια και στις ε, τροφές. Έτσι λοιπόν, χωρίς να ξανανοίγουμε τη συζήτηση για τη γλυφοζάτη, ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι έχει μείνει έχουν μείνει αρκετέ σοβαρέ ανησυχίε σε σχέση με την καρκο, καρκινογέννηση της ε, γλυφοζάτης. Από το 2015 από τη Διεθνή Οργάνωση Υγείας, το ίδιο για τη γλυφοζινάτη και ανεξάρτητες ε, μελέτες μας λένε, μας λένε ότι το ενεργό συστατικό 2,4D μπορεί να παραβλάψει το κυοφορούμενο και υπάρχουν και άλλοι ενδοκρινικοί διαταράκτες με σημαντικές συνέπειες για την υγεία. Η, η ζουξαφλουτόλη επίσης μπορεί να έχει πολύ σημαντικές ε, συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αξιολογήσεις επικινδυνότητας από την ΕΦΣΑ και έτσι δεν μπορούν τα προϊόντα αυτά να μπαίνουν ανεφετέρου στην τροφική αλυσίδα και τα τρόφιμα. Εμείς ως βουλευτές είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε και η διαδικασία πιστοποίησης των ε, γενετικά τροποποιημένων ε, οργανισμών που επεσήμανε και ο κύριος Γιούγκερ πρέπει να προχωρήσει προς περισσότερο εκδημοκρατισμό με τη διαδικασία της επιτροπολογίας την οποία περιμένουμε να δούμε να λειτουργεί με ένα σύστημα αξιόπιστο δημοκρατικό το οποίο όμως μέχρι να τεθεί σε ε, εφαρμογή θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι πολύ πιο αυστηρή ως προς τους ελέγχους και τις εγκρίσεις της. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενη μιλήτρια θα ήταν η κυρία Βερλίν που αντικαθίσταται ωστόσο από ε, την κυρία ε, Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ε, κυρία Χάσενκαμπ. Ε, όσα ήθελα να πω, τα είπε ήδη ο συνάδελφος, είναι πιστεύω σημαντικό να τονίσουμε ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της ε, Κομισιόν δεν συνάδει με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ούτε με το σκοπό και το στόχο του κανονισμού που βάσει των γενικών αρχών θέλει να παράσχει τη βάση για την παροχή υψηλής προστασίας ε, της ε, υγείας των ζώων και των ανθρώπων ε, και την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Ο κύριος λόγος για τον οποίο προβάλλουμε αντίρρηση έχει να κάνει με την γλυφοσάτη η οποία έχει καταταχθεί ως πιθανός καρκινογόνος προς τους ανθρώπους το Μάρτιο του 2015 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ε, και τη σχετική του επιτροπή και αυτή ο σοφασιόλος ο FG72 υποτίθεται ότι έχει ε, αντοχή στη γλυφοσάτη. Ε, εδώ μιλάμε για έλλειψη πρόληψης για την υγεία των ανθρώπων και έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της προφύλαξης. Επίσης η γλυφωσάτη εκκρεμεί επειδή η εξουσιοδότησή της ε, ε, λίγη τα του έτους. Οπότε πολλά έχουν πει ότι δεν πρόκειται να ε, ψηφίσουν υπέρ αυτής της ανανέωσης. Η δεύτερη κυρία αντίρρηση έχει να κάνει με τη διαδικασία. Από τότε που τέθηκε σε ισχύ η τρέχουσα εξουσιοδότηση, για τη γενικώς τροπημένη ουσία, οποιαδήποτε απόφαση έχει ληφθεί χωρίς ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών από την Κομισιόν. Και έτσι η εξαίρεση γίνεται ξαφνικά κανόνας. Κάτι το οποίο η, ε, η ίδια η Επιτροπή δεν βλέπει θετικά ως μη δημοκρατικό. Ε, κάθε φορά η Επιτροπή ΕΝΒΗ και η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, λένε ότι υπάρχει πρόβλημα στη διαδικασία. Αυτό θα πρέπει να γίνεται δίδαγμα και όχι να λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις. Ευχαριστούμε κυρία Εύη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να μιλήσω ως ε, συνυπογράφουσα αυτής ε, της αντίρρησης. Ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, που μίλησαν, παρουσίασαν όλοι στις αιτιολογίες που κάθε φορά μας οθούν να προβάλλουμε αντίρρηση στις νέες άδειε για προϊόντα γενετικώς τροποποιημένα εκ μέρου της Κομισιόν. Εγώ δεν ήθελα να επαναλάβω τα ίδια. Απλά να ρωτήσω την Κομισιόν δεν προτίθεστε να προβάλλετε μια νέα πρόταση ε, σε αντικατάσταση αυτής που απορρίφθηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε σχέση με την ε, ε, θέση στο εμπόριο των προϊόντων. Και μήπως θα ήταν σκόπιμο να αλλάξουμε τους κανόνες επιτροπολογίας Αφού γνωρίζουμε ότι μια τροποποίηση στον τεχνικό, τεχνικό κανονισμό για τα φυτά, τα ζώα και τη χορτονομή και τις ε, ζωοτροφές ε, θα μπορούσε να ευθυγραμμιστεί με τη, ε, όσα λέει η Τεχνική Επιτροπή για τα μηχανοκίνητα οχήματα όπου απουσία ειδική πλειοψηφία εντό της Τεχνικής Επιτροπής η Κομισιόν δεν μπορεί να προχωρήσει σε κάποια απόφαση ή άδεια Λαμβάνετε λοιπόν υπόψη αυτά τα στοιχεία ώστε να γίνει πιο δημοκρατική αυτή η διαδικασία αδειοδότησης των ε, γενετικώς τροποποιημένων ουσιών που όπως γνωρίζουμε σήμερα δεν είναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπάρας δεν είναι εδώ. Πάμε στους σκιώδεις. Α, συγγνώμη. Νόμιζα ότι καθόσασταν από εδώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Λέω εκ μέρους των σοσιαλιστών. Με ενοχλεί ιδιαίτερα που βρισκόμαστε και σε μια τέτοια συζήτηση και συζητούμαστε συντηρήσεις για ένα τεράστιο ζήτημα πρέπει να εκπροσωπήσουμε εδώ τους Ευρωπαίους πολίτες. Είμαι Ευρωπαίος πολίτης. Τι μπορώ να απαντήσω όταν γυρίσω στη χώρα μου. Αν μου πούν ότι επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα, τη γενετική ε, τροποποιημένη σόγια και ακόμα χειρότερα τη γλυφοσάτη. Με όλα αυτά που έχουμε ακούσει για αυτά τα ε, χημικά, όταν γνωρίζουμε ότι έχει, ε, υπάρχουν στοιχεία επιστημονικά που δείχνουν ότι υπάρχει σχέση της γλυφοσάτης με την καρκινογένεση. Πρόκειται για μια συζήτηση η οποία γίνεται στο δημόσιο διάλογο με πολύ έντονο τρόπο ήδη. Πέραν από τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, πώς μπορούμε να απαντήσουμε σε όλες αυτές τις ανησυχίες. Παρόλα αυτά λοιπόν, παρόλες αυτές τις ανησυχίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Όχι απλώς πρέπει να αλλάξει λοιπόν η διαδικασία από τη συνάδελφη, αλλά πρέπει να ρωτηθούμε γιατί έχει περάσει τόσο πολύ καιρό από την αρχή τη θητεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένει ότι πρέπει να αλλάξει η κατάσταση και δεν έχει συμβεί τίποτα. Επιμένουμε λοιπόν ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι πρέπει να αλλάξει η διαδικασία για να καταλήξουμε σε έναν κανονισμό, σε μια διαδικασία αποτελεσματική και μετά να απαγορεύσουμε τη χρήση τέτοιων προϊόντων τα οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Δεν μπορώ να ε, επιτρέψω με την ψήφη μου κάτι το οποίο θα δημιουργήσει προβλήματα στο, στο περιβάλλον, στην υγεία των παιδιών μου φαντάζομαι ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη που έχουμε απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες. Σας ευχαριστούμε. Θα δώσω το λόγο εκ μέρους των σκιωδών. Στον κύριο Κίζεκα. Συνάδελφος δεν μπορούσε να παρευρεθεί σήμερα, επομένως θα κάνω κάποιες σχετικές ε, παρατηρήσεις για τα, για τα γενετικά τροποποιημένη σόγια. Το Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2017 εκδόθηκαν σχετικές ε, ε, γνωμοδοτήσεις. Η ε, Επιτροπή για τα Γενετικά Τροποποιημένα της ΕΦΣΑ έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτά τα προϊόντα είναι ασφαλή για τη δημόσια υγεία και για το περιβάλλον. Από το 2015 έχουν υποβληθεί 20 αντιρρήσει στο προσχέδιο έγκριση γενετικά τροποποιημένων προϊόντων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει έναν κανονισμό τον οποίο ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητείται από την ΕΦΣΑ να διεξάγει μια επιστημονική αξιολόγηση. αυτό έχει συμβεί. Εάν η ΕΦΣΑ λοιπόν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το γενετικά τροποποιημένο προϊόν αυτό είναι ασφαλές, θα πρέπει να ακολουθήσουμε την επιστημονική της γνωμοδότηση. Δεν είναι ορθό να προσπαθεί κανείς από την πίσω πόρτα ε, και υπονομεύοντας την επιστημονική γνώση της ΕΦΣΑ να σταματά οποιοδήποτε έγκριση γενικά τροποποιημένων προϊόντων. Προτείνω λοιπόν στους συναδέλφους να καταψηφίσουν αυτές τις αντιρρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γκιολή. Thank you very much. Um, σας ευχαριστώ. Άλλη μια φορά λοιπόν που σε αυτή την Επιτροπή συζητούμε για μια εφαρμοστική πράξη η οποία όπως εξήγησαν και οι συνάδελφοι που παρουσιάζουν τις αντιρρήσεις δεν έχουν ε, ορθή νομική υπόσταση. Δηλαδή για άλλη μια φορά προσπαθούμε να υποκαταστήσουμε το σύστημα της επιτροπολογίας. Ακούμε επίση συναδέλφους να λένε ότι θα πρέπει να αλλάξει το σύστημα που το επιθυμούν. έτσι ώστε να μπορούν να σταματήσουν αυτές τις εξουσιοδοτήσεις. Ε, προσωπικά πιστεύω ότι είναι καλύτερα να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί εάν τεθείτε ενώπιον των ευθυνών σας και αν οι ψηφοφόροι σας γνωρίζουν ότι ήσασταν εσεί που σταματήσατε τέτοιου τύπου εξουσιοδοτήσει, ίσω να ε, το σκέφτεστε πλέον δύο φορέ. Έχουμε το πιο αυστηρό σύστημα στον κόσμο όσον αφορά την εξουσιοδότηση γενετικά τροποποιημένων προϊόντων, με πολλέ δυνατότητε να ληφθούν υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα και μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι οποιοδήποτε γενικά τροποποιημένο ε, προϊόν εγκρίνεται έχει το ίδιο επίπεδο ασφάλεια με οποιοδήποτε άλλο έχουν ληφθεί σχετικέ αποφάσει να μην επιτρέπεται η καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων προϊόντων μέσω τη διαδικασία τη ε, συναπόφαση. Και αυτό, δεν είναι... αυτό μάλιστα. Όμω, αυτό που προσπαθούν εδώ να κάνουν οι συνάδελφοι που παρουσιάζουν τι αντιρρήσει είναι να ε, σταματήσουν την εξουσιοδότηση ενό προϊόντο το οποίο ήδη χρησιμοποιείται στι ΗΠΑ ε, στι ζωοτροφέ. Δεν πρόκειται για δεν έχω ακούσει μάλλον αντίστοιχε αντιρρήσει στην συζήτηση που είχαμε στον τον Ιούλιο. Είναι ξεκάθαρο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν επέτρεψε στα κράτη-μέλη να αποφασίζουν κατά τη διακριτική τους ευχαίρεια να χρησιμοποιούν ή όχι ε, αυτά τα προϊόντα για τις ζωοτροφές. Αυτό θα ήταν ένα πολύ δύσκολο θέμα γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει επάρκεια ε, στις, ε, στα προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ζωοτροφές. Συνεχίζοντας λοιπόν σε αυτόν τον δρόμο, με αυτό, σε αυτόν τον δρόμο, δεν θα καταφέρουμε ποτέ να είμαστε ε, αυτάρκης στον τομέα αυτών. Έχουμε εκστρατείες από τους ίδιους συναδέλφους κατά των βιοκτώνων, κατά των φυτοπροστατευτικών μέσων, οτιδήποτε δηλαδή θα μπορούσε να βοηθήσει στην παραγωγή ε, καλλιεργιών που θα οδηγούσε σε, σε, σε επάρκεια της, των ζωοτροφών, της παραγωγής ζωοτροφής. Ακολουθώντας το σκεπτικό τους, ε, δεν ε, υπάρχει καμία δυνατότητα για τεχνολογική καινοτομία. Αγνοούν τις επιστημονικές αναλύσεις οι ίδιοι συνάδελφοι διαμαρτύρονται όταν, αγνο, όταν αγνοούνται οι επιστημονικέ αναλύσει για την κλιματική αλλαγή. Όμω για αυτό το ζήτημα φαίνεται ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να αγνοούμε τα επιστημονικά δεδομένα. Δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν γιατί από πού και ως πού ακολουθούν τη, μια ιδεολογική βάση χωρίς κανένα επιστημονικό δεδομένο να τους υποστηρίζει. λένε ότι αυτά τα προϊόντα ε, χρησιμοποιούνται χωρίς καμία εξουσιοδότηση. Είναι στον αέρα. Δεν είναι καθόλου στον αέρα. Υπάρχουν οι ίδιες ε, ε, αυστηρές εξουσιοδοτήσεις που χρησιμοποιούνται και για οποιοδήποτε που υποβάλλονται και για οποιοδήποτε άλλο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να καταψηφιστούν αυτές οι αντιρρήσεις. Δυστυχώς φοβάμαι που δεν θα συμβεί αυτό. Αλλά όπως είπα Προσβλέπω στην ημέρα όπου θα λογοδοτείτε για αυτές τις αποφάσεις σας να μην επιτρέπετε την εξουσιοδότηση τέτοιων προϊόντων αγνοώντας τα επιστημονικά δεδομένα. Σας ευχαριστούμε. Εκπρόσωπος της Επιτροπής, ο κ. Μπέρντ. Thank you very much, Madam Chair. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, ευχαριστώ για τα σχολεία σας και ευχαριστώ που δένετε τη δυνατότητα στην Κομισιόν να ε, σχολιάσει αυτά τα δύο σχέδια ψηφίσματος. Ζητώ συγγνώμη από τον συναδελφό μου που δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ σήμερα και μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω. Να τονίσω πρώτα απ' όλα ότι αυτές οι δύο αιτήσει όσον αφορά την έγκριση φασιολουσόγιας ε, για ε, ζωοτροφές δεν αφορά την καλλιέργεια. Αυτό το είπε πολύ σωστά η κυρία Γκέρλεγκ στην παρέμβασή της και η Κομισιόν έχει ακολουθήσει όλα τα διαδικαστικά βήματα που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία για τα γενετικώ τροποποιημένα. Η ΕΦΣΑ πραγματοποίησε την αξιολόγηση των προϊόντων με θετικά συμπεράσματα και για τα δύο γενετικώ τροποποιημένα προϊόντα, με θετικέ ε, επιπτώσεις για τα ζώα και για το περιβάλλον. Ε, τα, σχόλια, τα κρατημέλη σχολίασαν αυτή την εκτίμηση ε, επικινδυνότητας και η ΕΦΣΑ σχολίασε τα σχόλια αυτά στην ε, σχετική συνάντηση. Δεν υπήρξαν σχόλια από τα κράτη-μέλη κατά της θετικής γνωμοδότησης της ΕΦΣΑ και το κοινό σχολίωσε ε, τις γνωμοδοτήσεις της ΕΦΣΑ στα οποία σχόλια απάντησε η ΕΦΣΑ είναι θετικές οι γνωμοδοτήσεις για αυτή τη σόγια. Βάσει των παραπάνω, η Κομισιόν πρότεινε στα κράτη-μέλη να αδειοδοτήσουν αυτούς τους βασιλούς σόγιας δυνάμει του κανονισμού 8029 του 2003 και της Γενικής Νομοθεσίας Περιτροφίμων. Όπως περιγράφει και ήδη από δύο αξιότιμα μέλη, οι αποφάσεις ψηφίστηκαν τον Ιούλιο του 2017, χωρίς ε, ειδική πλειοψηφία κατά υπέρ, ε, κυρίως λόγω πολιτικών λόγων και της αρνητικής κοινή γνώμης και όχι για λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με τους κανόνες ε, επιτροπολογίας, και με τον κανονισμό ε, για τις ζωοτροφές ε, και τη χορτονομή. 14 ε, Σεπτεμβρίου 2017 παρουσίασε την πρόταση Κομισιόν χωρίς να υπάρχει αποτέλεσμα κάποια γνωμοδότηση όσον αφορά τα σχόλια του σχεδίου κανονισμού κατά την άψη της Κομισιόν η προσέγγιση πολιτικής δεν παρουσιάζει πρόβλημα η απόφαση να επιτραπεί σε μια τρίτη χώρα η καλλιέργεια γενετικώ τροποποιημένων προϊόντων είναι απόφαση της εν λόγω χώρο. Δεύτερον, πρέπει να θυμόμαστε ότι όταν εισάγουμε τρόφιμα ε, και ζωοτροφές από μια τρίτη χώρα εξακολουθούν να ισχύουν τα πρότυπα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και όλες οι χώρες ε, ε, συμμετέχουν στο Διεθνέ Πρωτόκολλο Ασφαλείας. Οι ΙΠΑ έπαιξαν ενεργό ρόλο σε όλη τη διαδικασία για τη συμφωνία των ε, στόχων βιώσιμη ανάπτυξη και για το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και του σχετικού στόχου εντό Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την αναπτυξιακή συνεργασία με τι χώρε εταίρου. Όσον αφορά το θέμα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, και το θέμα της γλυφοσάτης που αναφέρθηκε πολλές φορές ε, στην οποία έχουν αντοχή τα, οι φασιολισόγειας όπως για όλες τις καλλιέργειες αυτά τα γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα όταν εισάγονται πρέπει να συμμορφώνονται με τα μέγιστα επίπεδα καταλήπων που ορίζονται σε ξεχωριστή νομοθεσία και που δεν ρυθμίζονται από τον κανονισμό για τα γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα. Παρομοίω, ε, η, έγκριση, η ανανέωση τη έγκριση για τη γλυφοσάτη δεν ρυθμίζεται από τον κανονισμό για τα γενετικώς προϊόντα και όπω ανέφερε η κυρία Γκέρλινγκ η συζήτηση για την ανανέωση. Αυτή, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη πράγματι και οι απόψει των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ΕΚΑ και ΕΦΣΑ, ε, διαφέρουν από αυτό που αναφέρει η κυρία Χάζεκαμπ ε, στην ομιλία της. Επίσης, ο σχεδιασμός των δοκιμών περιλάμβανε τον ψεκασμό της σόγιας με καθένα από τα εν λόγω και με όλα τα ζενοκτώνα μαζί και όπως φαίνεται, όπως λέει η Κομισιόν, υπήρξε τήρηση των προτύπων ε, που προβλέπει η ΕΦΣΑ, έγιναν ψεκασμοί σωστά. Όσον αφορά την έκκληση για αναστολή αυτών των σχεδίων αποφάσεων ε, ως την αναθεώρηση της ε, απόφαση αδειοδότηση. Ε, να υπενθυμίσω ότι η Κομισιόν έχει υποβάλει πρόταση που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να περιορίσουν τι εισαγωγέ γενετικώ τροποποιημένων ε, τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά του. Δυστυχώ αυτή η πρόταση απορρίφθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ενώ αναμένουμε να δούμε τι συζητήσει στο Συμβούλιο για την πρόταση αυτή. Επιπλέον, για να απαντήσω σε μια από τι ερωτήσει τη κυρία Εύη η Κομισιόν επίση έκανε μια πρόταση τροποποίηση των κανόνων που διέπουν την διαδικασία επιτροπολογία. γεγονός που θα δώσει μεγαλύτερη ευθύνη στα κράτη-μέλη. Η πρόταση αυτή συζητείται αυτή τη στιγμή από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Εώσο ότου όμως ολοκληρωθεί αυτή η νομοθετική διαδικασία, η υπάρχουσα διαδικασία εξακολουθεί να ισχύει. Και αυτό πρέπει να το σεβαστεί η Κομισιόν. Συμπερασματικά να υπογραμμίσω ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο να αποσύρει η Κομισιόν αυτό το σχέδιο αποφάσεων να που αφορούν την εξοδότηση εισόδου στην αγορά αυτών ε, των φασιολών σόγια. σόγια βάσει των αποφάσεων τη ΕΦΣΑ έχουν ακολουθηθεί όλε οι προβλεπόμενε διαδικασίε στην νομοθεσία και η Κομισιόν ε, δρά αυστηρά εντό των εκτελεστικών τη αρμοδιοτήτων. Να πω επίση ότι το δικαίωμα εξέταση του ε, ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιορίζεται στο ζήτημα του κατά πόσο υπερβαίνει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται για την εκτελεστική πράξη και η Κομισιόν ε, τονίζει ότι δεν έχει ε, λάβει χώρα τέτοια υπέρβαση, δεν μπορεί να ελέγξει το σχέδιο απόφαση για άλλα θέματα που αναφέρονται στην αντίρρηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζω οι εξηγήσει που έδωσα να απαντούν στα σημεία που ε, αναφέρονται στο σχέδιο αντίρρηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και έτσι ολοκληρώνεται η πρώτη συζήτηση για αντίρρηση σήμερα. Για να δούμε και τη δεύτερη. Ακριλομίδη. Ο κύριος Κάρας αντικαθιστά την ε, συντάκτρια. Παρακαλώ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η κυρία Κωστινγκέρ με παρακάλεσε να σας συγγνώμη εκ μέρου τη και να παρουσιάσω εν συντομία το θέμα που την ενδιαφέρει. Έχουμε λοιπόν την αντίρρηση για την νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για τη χρήση μέτρων ελέγχου και περιορισμού για την μείωση του περιεχομένου σε τρόφιμα της σε ακριλαμίδη. Πιστεύω ότι όλοι θα πρέπει να συμφωνούμε πως οτιδήποτε έχει καρκινογόνες συνέπειες και υπάρχουν σχετικές αποδείξεις ότι μπορεί να έχει καρκινογόνες συνέπειες η ακριλαμίδη, πρέπει και οφείλει η Επιτροπή αντίστοιχα να μεριμνήσει για την προστασία της υγείας των πολιτών. Πρέπει λοιπόν να ελέγχονται αυστηρότερα για να μειώνεται στο δυνατόν ο κίνδυνος. Έτσι λοιπόν, με την αντίρρηση αυτή δεν είναι τίφτε ζήτημα προστατεύουμε νέου, αλλά ξεκαθαρίζουμε το ζήτημα, προστατεύουμε ναι και τελεία. Εδώ λοιπόν μας έχει προκύψει ε, το ζήτημα λόγω της αβεβαιότητας ως προς την εφαρμογή του κανονισμού, κατά, ως προς την ε, διεξαγωγή των ελέγχων κατά την εφαρμογή του κανονισμού, γιατί υπάρχει ένας ε, μακροσκελέστατος ε, κατάλογος μέτρων που καταγράφεται ε, και που οδηγεί σε υπερβολική γραφειοκρατική επιβάρυνση της, του κλάδου της σύντησης και των εστιατορίων και της εστίασης και ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί η ίδια ότι θα πρέπει να προταθούν κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες θα διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να προβαίνουν σε αυτές τις ε, διατυπώσεις τις γραφειοκρατικές και πώς μπορούν να απαλλαγούν από τον υπερβολικό φόρτο. Γι' αυτό λοιπόν συζητούμε και τις συνέπειες του κανονισμού ώστε να αποφύγουμε την υπερβολική αβεβαιότητα που θα μπορούσε με τη σειρά της να οδηγήσει σε ε, επιθέσεις άδικες εις βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα από τις τηγανιτές πατάτες. Πρέπει, λέει, ή δυνατόν οι τηγανιτές πατάτες ε, πριν τηγανιστούν να έχουν πληθεί και να έχουν μείνει περίπου 30 λεπτά σε νερό και ούτω καθεξής εδώ στην Αυστρία. Έχουμε να κάνουμε με μάγειρες, με ανθρώπους όπου, ε, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει ε, πρακτική εξάσκηση, μαθήματα, κατάρτιση. Είναι άνθρωποι εξειδικευμένοι. Και γι' αυτό λοιπόν κάνουμε μία πρόταση για να γίνει σεβαστή και η δουλειά που κάνουν αυτοί οι επιχειρηματίες και να μην επιβαρύνονται υπερβολικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλες αυτές τις οδηγίες και διατάξεις. Κάνουμε την πρόταση λοιπόν μιας εξαίρεσης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και λέμε και πάλι πως όντως πρέπει να γίνει παραπομπή στην σύσταση του 2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο τη βελτίωση της δημόσιας υγείας που όμως δεν μας ε, εξασφαλίζεται πιστεύουμε γιατί δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Το θέμα δεν είναι να κάνουμε κάτι δηλαδή αλλά να φέρουμε και πάλι στη συζήτηση τη δυνατότητα για απλοποίηση των κανόνων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατ' εξαίρεση για λόγους ασφάλειας δικαίου και βέβαια αντίστοιχα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει μόνο έναν καθοδηγητικό ρόλο. για να μην αναλαμβάνουν δραστηριότητες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χωρίς να γνωρίζουν ποιοι είναι οι κανόνες. Έτσι λοιπόν θέλουμε με την πρόταση της κυρίας Κιόσνιγκερ που υποστηρίζουμε μια απλοποίηση, μια απλούστευση των κανόνων. Σας ευχαριστώ πολύ και εκ μέρους ομάδας μου βεβαίως για την υποστήριξη αυτού της αντίρρησης. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μίλοχ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Είχαμε πριν το καλοκαίρι στη Γερμανία ε, μεγάλη φασαρία που ξέσπασε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται να ε, επιβάλλει ρυθμίσεις και στις τηγανικές, τηγανιτές πατάτες. Και χρειάστηκε βέβαια να κάνουν τι σχετικέ ανακοινώσει και απαντήσει φαντάζομαι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, για να καθισχύσουμε του πολίτε. Εάν η πρόταση, αν κοιτάξει κανεί την πρόταση για τα μέτρα ελέγχου ή περιορισμού των ποσοτήτων ακριλαμίδη, νομίζω θα καταλάβει περί τίνο πρόκειται. Όταν πρόκειται για μικρέ μεσές επιχειρήσει και παραγωγέ, θα πρέπει να έχουμε διαφορετικέ προσεγγίσει, γιατί είναι μικρέ και πολύ μικρέ επιχειρήσει, οι οποίε κινδυνεύουν να μην μπορούν να κάνουν τη δουλειά του με επάρκεια ε, λόγω αυτών των γραφειοκρατικών επιβαρύσεων. Και τις τελευταίες εβδομάδες καταβάλαμε μεγάλες προσπάθειες με πολλές συζητήσεις σε συνεργασία κυρίως με τους εκπροσώπους των εμπλεκομένων ε, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, από τις οποίες συζητήσει προκύπτει για μένα ξεκάθαρα το γεγονός ότι μετά την συζήτηση και το πλαίσιο μιας βελτιωμένης νομοθεσίας θα έχουμε καλύτερη προστασία των καταναλωτών χωρίς να υποχρεώσουμε τις ε, επιχειρήσεις αυτές να αλλάξουν τα προϊόντα τους ή να τις επιβαρύνουμε με υπερβολικό γραφειοκρατικό φόρτο. Η υποστήριξη των διαφόρων ομάδων συμφερόντων ε, για την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκφράζεται σε ευρύ φάσμα στη Γερμανία και έτσι την αντίρρηση εμείς ε, θα είχαμε τάση μάλλον να την απορρίψουμε. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αμελήσουμε ή να λησμονήσουμε, δεν σας το κρύβω αυτό, ότι πρέπει να υπαγρυπνούμε ε, και να διαρωτόμαστε τι πραγματικά μπορεί να έχει γίνει λάθος ως προς την επικοινωνιακή μας πολιτική, τι πηγαίνει στραβά ως προς την επικοινωνιακή πολιτική, γιατί όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν ε, χωρίς ε, αποτέλεσμα εκεί που κάναμε συζητήσεις ανόητες για, την, ε, για το τουρσί αγκουράκι ή αγκούρι λαχανικό έχουν πάει χαμένα και νομίζω ότι θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε για κάτι πιο ουσιαστικό. Κύριο Στέιλορ. Well, thanks very much, Chair. Um, well... Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα τις δύο συναδέλφους και την Και θα ήθελα να διαβεβαιώσω στους συναδέλφους ότι κανείς δεν αμφιβάλλει για το, τις των μαγείρων στην Αυστρία. Αυτό που μας ανησυχεί είναι ο κίνδυνος ε, από αυτά τα τρόφιμα από ένα πιθανό λάθος. Θα ήθελα να ξεκαθαρίζω ότι διαφωνούμε με το να αναβληθεί η ψηφοφορία για αυτές τις αντιρρήσεις, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει λόγος. Επίσης να σας πω ότι θα καταψηφίσουμε τις αντιρρήσεις για τους εξή λόγου. Το 2015 η Επιτροπή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η ΕΦΣΑ, εξέδωσε γνωμοδότηση η οποία επιβεβαίωσε προηγούμενες γνωμοδοτήσει τη ότι το ακριλαμίδιο στα τρόφιμα είναι πιθανόν να αυξήσει, αυξάνει μάλλον την πιθανότητα καρκινογένεσης. Όμως, ο της ποσότητας του ακριλαμίδιου στα τρόφιμα ε, για όλες τις ηλικιακές ομάδες ε, καταδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος καρκινογένεσης. Και ευτυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε δράση μετά από αυτή τη γνωμοδότηση με πρόταση ε, για την μείωση του ποσοστού ακριλαμιδίου στα τρόφιμα που την οποία πρόταση θα πρέπει να τηρήσουν όλοι, όλες οι επιχειρήσεις. Τα κατόφλια λοιπόν, τα οποία καθορίζονται στην νομοθεσία, δεν είναι υψηλά. Το 85 με 90% των τροφίμων που βρίσκονται στην αγορά ήδη τα τηρούν. Άρα, σε αντίθεση με αυτά που λέει η συνάδελφος Κέστινγκ, δεν θα δημιουργηθεί τεράστιο άχθος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή για οποιαδήποτε επιχείρηση, οι οποίες έτσι και αλλιώ γνωρίζουν, ότι έχουν ευθύνε όταν θέτουν οποιοδήποτε τρόφιμα στην αγορά. Αντιθέτω, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, του κλάδου της εστίασης, οι ε, απαιτήσει είναι ακόμα λιγότερο δυσβάσταχτες. Ε, Η πρόταση της Επιτροπής προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τους δραστηριοποιούμενους στον κλάδο των τροφίμων για τους κινδύνους του ακριλαμιδίου. Σας ζητώ λοιπόν, τη συνάδελφοι, να καταψηφίσετε αυτές τις αντιρρήσεις. Κυρία Σάντελ, λοιπόν, των Σοσιαλιστών. Υποστηρίζουμε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό θα καταψηφίσουμε τι αντιρρήσει που έχει υποβάλει το ΕΛΚ. Για του εξή λόγου. Το πρώτο μα μέλημα είναι η προστασία τη υγεία των καταναλωτών στην Ευρώπη. Το 2015, όπω είπε και ο συνάδελφο, η ΕΦΣΑ έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, είπε ότι τα επίπεδα κρυλαμιδίου στα τρόφιμα είναι εξαιρετικά υψηλά. Και προσπαθούμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Ακούμε το ΕΛΚ να μας λέει ότι αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επειδή δημιουργεί γραφειοκρατία. Ε, όμως αυτό δεν ισχύει. Από την τις γνώσεις που αποκόμισα, από τα μήνυματα που έλαβα από διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, από εκπροσώπους του κλάδου, Για παράδειγμα, η Food Drink Europe ε, μας αναφέρει ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ρεαλιστική και δίκαιη και εύκολο να εφαρμοστεί πρακτικά. Ε, για την αντιμετώπιση του προβλήματος του ακριλαμιδίου. Κάτι αντίστοιχο λένε και οι Αρτοποιοί. Ε, υποστηρίζουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηλαδή. Αν λοιπόν κάποιο ήθελε να ασκήσει κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό που θα έπρεπε να τις προσάψουμε είναι ότι δεν, έγινε, δεν έλαβε ακόμα πιο αυστηρές πρωτοβουλίες για τον περιορισμό του ακριλαμιδίου. Η ομάδα των σοσιαλιστών λοιπόν υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για το ακριλαμίδιο και θα καταψηφίσει τις αντιρρήσεις του ΕΛΚ. Θεωρούμε ότι η πρόταση που μας υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εύλογη και δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στον κλάδο. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω, είναι μεγάλος ο κατάλογος. Ήμουν βέβαια ότι θα συνέβαινε αυτό και έχουμε και άλλη μια αντίρρηση που πιστεύω ότι θα προκαλέσει το ίδιο πολλέ αντιδράσει και θα πρέπει να τι συζητήσουμε πριν από την ψηφοφορία, διότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε χωρί ε, συζήτηση. Οπότε έχετε το υπόψη σα όταν μιλάτε ή όταν σηκώνετε το χέρι σα, παρουσιάστε επιχειρήματα που δεν έχουμε ακούσει από του προηγούμενου ομιλητέ, αν είναι δυνατόν. Επόμενο ομιλητή, ε, κύριο Λίσα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Το κρυλομίδιο είναι βεβαίως πρόβλημα για την δημόσια υγεία. παίρνουμε δείγματα από νέους και εγώ ως ε, γιατρός έχω διαπιστώσει αυτό το πράγμα στις συνομιλίες μου με τους ειδικού. πολιτικά. Ωστόσο, σημειώνω και επιπλέον σημειώνω ότι ο κίνδυνος προκύπτει από, την, από το ακριλαμίδιο στην Ευρώπη είναι μεγαλύτερος από αυτόν της γλυφοζάτης και των λοιπών. Πρέπει λοιπόν γι' αυτό να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Και το λέω και για όλους τους δημοσιογράφους που ενδεχομένως παρακολουθούν τη συζήτηση αυτή και στην Αυστρία και στη Γερμανία, την Bild και άλλες εφημερίδες που έχουν προβάλει το θέμα αυτό. Είναι ε, ο κίνδυνος τέτοιο πρέπει να ενημερώνονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γιατί δυστυχώς Το μεγαλύτερο κίνδυνο από ακριλαμίδιο τον, τον ε, προξενούμε εμείς οι ίδιοι από τις τροφές που ετοιμάζουμε στο σπίτι μας, από το ψωμί το οποίο βάζουμε στην τοστιέρα, από την πατάτα που τηγανίζουμε στο δικό μας τηγάνι και καίγεται. Αυτός λοιπόν ο μεγαλύτερος κίνδυνος και αυτό πρέπει με την ε, σωστή πληροφόρηση Ε, πρέπει με τη σωστή πληροφόρηση λοιπόν και ενημέρωση να το καταστήσουμε γνωστό στο κοινό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί με αρελισμό την ε, κατάσταση με τη σωστή προσέγγιση κατά, τη θέση, κατά τις θέσεις μας, αλλά η κατάσταση είναι δύσκολη και για τον εξή λόγο, διότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακολουθεί μεν μια συγκεκριμένη προσέγγιση, αλλά όχι τόσο σαφή, δηλαδή αφήνει περιθώριο για πολλές διαφορετικές πληροφορίες ή συμπεράσματα και έτσι οι εκπρόσωποι του κλάδου μας λένε καλή, καλός ο δρόμος που έχετε πάρει, θέλουμε και πιο σαφείς ε, οδηγίες. Τώρα από πρώτου του 2018 πρόκειται να θέσει σε εφαρμογή χωρίς όμως σε γραμμές αυτό το μέτρο. Α ξεκινήσει λοιπόν η διατύπωση των κατευθυντικών γραμμών το ταχύτερο δυνατό, ώστε να κλείσει το θέμα αυτό, αλλά η κατάσταση είναι αυτή που μα περιέγραψε και ο Τμαρκάρας, ότι εάν αφήσουμε τώρα να μα ξεφύγει από τα χέρια αυτή η κατάσταση, δεν έχουμε κανένα τρόπο να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να διευκρινίσει την κατάσταση γι' αυτό και θέλουμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ταχύτερο δυνατόν και όχι γενική διεύθυνση όχι μέσω της Γενικής Διεθνής, αλλά με απόφαση της Επιτροπής ως συλλογικού οργάνου ε, να προβεί σε μια διευκρίνηση κατάστασης και να μην περιμένει βέβαια την 1η Ιανουαρίου γι' αυτό. Δύο συγκεκριμένα είναι τα αιτήματα των εμπλεκομένων και ενδιαφερομένων φορέων. Πρώτον, διευκρίνηση της νομοθεσίας. Δύο-τρία, τμήματα δύο-τρία και τρία του δεύτερου παραρτήματος, ε, θα πρέπει να ισχύουν μόνο για τις μεγάλες αλυσίδες εστιατορίων και το τμήμα Α του δεύτερου παραρτήματος να διευκρινιστεί ότι αφορά μόνο σύσταση και όχι υποχρέωση. Εγώ έτσι θεωρώ ότι ισχύει, αλλά δεν μπορεί κανείς να είναι βέβαιος. Και μια και υπολείπονται μόνο μερικές εβδομάδες να τεθεί σε εφαρμογή. Καλό θα είναι να εξεταστεί από την Επιτροπή ε, στην συλλογική της σύνθεση η υπόθεση αυτή για να διευκρινιστεί με απόλυτη σαφήνεια. Υποστηρίζουμε λοιπόν την πρόταση, αλλά ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε ταχύτερα σε μια συμφωνία ώστε να δοθούν οι διευκρινήσεις εγκαίρως. Για τον λόγο αυτόν και πρώτον επειδή θέλουμε αυτήν την συμφωνία αλλά και δεύτερον γιατί θεωρούμε ότι πρέπει η Επιτροπή ως λογικό όργανο να το εγκρίνει το θέμα παρακαλούμε να αναβληθεί η αντίρρηση αυτή ωστόσο ζητούμε από τους συναδέλφους ε, να λάβουν ε, υπόψη ε, ότι σήμερα έχουμε όλη τη μέρα η μερίδα εργασία ω ΕΛΚ στη Ρώμη. Δεν θα είναι δυνατόν δηλαδή να είναι όλοι παρόντε στην ψηφοφορία. Ε, γι' αυτό παρακαλούμε και για την αναβολή. Έχουμε χρόνο όμω, εάν το προβλέψουμε για την προσεχή μα συνεδρίαση, προσεχή συνεδρίαση τη Επιτροπή, να κάνουμε ψηφοφορία εκεί. Η Πρόεδρο. Να ζητήσω να μην μακρηγορείτε, α μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια, διότι τα έχουμε ακούσει πολλέ φορέ και απομπαίνουν πολλά πρέπει να κάνουμε. Κυρία Γκέρλινγκ, ε, ζητώ συγγνώμη που είστε επόμενοι συνήθω. Ε, τηρείτε του χρόνου θα σας πάρω πολύ σοβαρά και θα περιοριστώ σε λίγα λόγια. Δεν θα υποστηρίξω την αντίρρηση. Μίλησα νωρίτερα για την επιστημονική συνένεση. Είναι σαφώς ότι, σαφώς ότι υπάρχει συνένεση ότι το ακριλαμίδιο αποτελεί απειλή για την υγεία. Η πρόταση αυτή είναι μια σωστή προσέγγιση. Κάτι που με ανησυχεί ειδικότερα είναι οι αρνητικές επιπτώσεις για τις μικρές επιχειρήσεις. Το εξετάσαμε προσεκτικά εξετάσαμε την υποχρέωση της Κομισιόν ε, προς τις μικρές επιχειρήσεις και πιστεύουμε ότι πλήρηται. Και έχουν προβλεφθεί κάποιες εξαιρέσεις που θα βοηθήσουν τις ε, ε, μικρές επιχειρήσεις, οπότε θα υποστηρίξουμε την αντίρρηση. Ευχαριστούμε, κύριε Σπεντιτσίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να υπενθυμίσω στο ΕΛΚΑ ότι οι πιο μεγάλες ομάδες ε, τροφίμων που ε, έχουν ακριλαμίδι αφορούν τα παιδιά. Την πιο ευαίσθητη ηλικία σε τέτοιου είδους έκθεση. Οπότε μας κάνει έκπληξη αυτή η χιλιοστή προσπάθεια καθυστέρησης ε, της υιοθέτησης αυτών των εκτελεστικών μέτρων. Να υπενθυμίσουμε ότι από το 2005 όταν η ΦΑΟ συμπέρανε ότι τα επίπεδα έκθεση στο ακριλαμίδιο ε, αποτελούσαν συναγερμό για την ανθρώπινη υγεία και το 2015 η ΕΦΣΑ επανέλαβε ότι η παρουσία κρυλαμιδίου στα τρόφιμα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου για καταναλωτές πάσης ηλικία. Οπότε έχουμε καθυστερήσει σημαντικά στην έγκριση αυτού του πράγματος ε, και το επενθυμίζω στο ΕΛΚΑ. Ε, εδώ δεν ορίζονται δεσμευτικά όρια, μόνο κάποια όρια εθελοντικά, ελαφρά όρια για τις εμπορικές δραστηριότητες ε, μικρής εμβέλειας ε, δεν θα επηρεάσει κανένα παραδοσιακό ε, φαγητό. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν τι σας ανησυχεί για μας. Η πρόταση της Κομισιόν να πρέπει να εγκριθεί αμέσω. Αποτελεί για μας μόνο μια αφετηρία για μια μεγαλύτερη διαδρομή ευρύτερης προστασίας της ανθρωπινής υγείας. Ευχαριστούμε κυρία Κονέτσνα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω εκ μέρους της ομάδας μου. Εμείς θα ψηφίσουμε κατά της πρότασης φυσικά. Και θα ήθελα να σας ζητήσω να μην αναβάλλετε την ψηφοφορία, διότι ακούγοντας τον κύριο Λίζερ το να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε όλα μας τα έγγραφα για την Κομισιόν, αυτό θα ήταν επιχείρημα κατά ημών, αν το αφήσουμε να εκκρεμεί. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιο κατά ημών. Οι εμπειρογνώμονες συμφωνούν ότι η γνωμοδότησή τη ΕΦΣΑ ε, κυκλοφόρησε πριν από δύο χρόνια. Σύμφωνα με αυτή την γνωμοδότηση λοιπόν είναι καρκινογόνο το ακριλαμίδιο και όλοι οι εμπειρογνώμονες όλων των κρατών μελών ε, συμφωνούν από αυτού. Δεν βλέπω λοιπόν να υπάρχει λόγος για αναβολή τη ε, θέση σε ισχύ Η Κομισιόν θα μπορούσε να έχει εκδώσει βέβαια κατευθύντηρε γραμμέ, αλλά αν ε, πραγματοποιήσουμε αναβολή ενό μήνα ε, περίπου, θα κολλήσει φοβάμαι κάπου και θα οδηγηθούμε σε βεβαιότητα. Η ομάδα ε, της GUE-NGL δεν ξεχνά ποτέ την προστασία των καταναλωτών. Αποτελεί κομμάτι του πολιτικού μας προγράμματος ε, το έχουμε προβάλει και στα κράτη-μέλη μας. Ε, το να απορριφθεί λοιπόν αυτή η αντίρρηση είναι προτεραιότητα για μας σήμερα. Δεν πρέπει να διστάζουμε άλλο. Ευχαριστούμε κύριε Κάμπαχ. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν σαφή νομίζω οι τοποθετήσεις. Είναι σαφέ ότι όλοι οι περισσότεροι εδώ θεωρούν ότι είναι επικίνδυνο για την, επικίνδυνο για την υγεία το άκρη λαμίδιου. Πρέπει νομίζω να οργανώσουμε να ε, υποστηρίξουμε την ε, πρόταση που έχει οθετήσει και προβάλλει ως αντίρρηση αυτή η συνάδελφος η οποία αποχωρεί για να αναλάβει καθήκοντα στην Αυστρία. Ε, πρόκειται για μία ιδέα την οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποστηρίζει ο Ότμαρ Κάρα. Πρέπει να υπάρχουν κατευθυντήριε γραμμέ, συστάσει, διευκολύνσει για τι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει. Είναι δεδομένα λοιπόν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, δεν χρειάζεται τίποτε περισσότερο. Πρέπει λοιπόν να απορριφθεί ε, και η αναβολή και το αίτημα τη κυρία Κρίστιγκερ. Commission, Mr. εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Όπως αναφέρθηκε ήδη, πράγματι η ΕΦΣΑ έκανε μια εξαντλητική επιστημονική γνωμοδότηση το 2015, στην οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι για όλες τις ηλικιακές ομάδες το ποσοστό ακριλαμιδίου στο οποίο εκτίθενται ε, δημιουργεί κινδύνους για την εμφάνιση καρκίνου. Ήδη από το 2002 εντοπίστηκαν ποσότητες ακριλαμιδίου στα τρόφιμα. Και έχουν γίνει πολλά από τότε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. αναφέρεται το θέμα στην έκθεσή μας το 2014. Και εκτός αυτού, ήδη ο κλάδος έχει αρχίσει να προσπαθεί να αναπτύσσει εργαλεία για τον περιορισμό του ποσοστό του ακριλαμιδίου ε, που χρησιμοποιούνται σε θελοντική βάση. Ωστόσο, από την διερεύνηση του προβλήματος που επί τη βάση της ίστασης Επιτροπής έκαναν τα κράτη-μέλη, φαίνεται ότι αυτά τα εθελοντικά μέτρα περιορισμού ε, της χρήσης ακριλαμιδίου, της, της, της εμφάνισης ακριλαμιδίου στα τρόφιμα, ε, εφαρμόζονταν με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με την επιχείρηση ε, που δραστηριοποιείται στον κλάδο των τροφίμων και ε, αυτή η κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική. Αυτό που σας είπα το επιβεβαιώνει και η γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ του 2015, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν διαφορές και δεν έχει μειωθεί συστηματικά το κρυλαμίδιο στα τρόφιμα τα τελευταία χρόνια. Για αυτούς τους λόγους κατέληξε στο συμπέρασμα η Επιτροπή ότι χρειάζονται ρυθμιστικά μέτρα για να μειωθεί το ακριλαμίδιο και ε, για να καταστούν υποχρεωτικά αυτά τα μέτρα περιορισμού του ακριλαμίδιου για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Κάνοντας όμως αυτά τα μέτρα υποχρεωτικά, η Επιτροπή φρόντισε ε, να τα προσαρμόσει ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των εστιατορίων, των περιπτέρων που πουλάνε τριτηγανιτές πατάτες. Για παράδειγμα, υπάρχουν ρητές εξαιρέσεις ε, που απο... Ε, προβλέπουν ότι δεν χρειάζεται μια μικρομεσαία επιχείρηση να κάνει δειγματοληψία ή να τηρεί αρχεία. Φροντίσαμε να μην δημιουργηθεί λοιπόν επιπλέον επιβάρυνση γραφειοκρατικού χαρακτήρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το προσχέδιο κανονισμού έχει εξεταστεί εκτενώς το τελευταίο 1,5 χρόνο από εκπροσώπους του κλάδου και επαγγελματίες του χώρου, της εστίασης, ε, διαφόρων μεγεθών. Δημοσιοποιήθηκε επίσης στο, στην πύλη για το ευνομοθετήν το Better Regulation Portal της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Λάβαμε πολλά σχόλια τα οποία τα εξετάσαμε ενδελεχώς και αυτά τα σχόλια οδήγησαν και σε αλλαγές στο προσχέδιο του κανονισμού πριν αυτό ε, το προσχέδιο υποβληθεί προς ψήφιση τον Ιούλιο στην Διαρκή Επιτροπή για την ασφάλεια των τροφίμων. Όμως, όπως ο κύριος Λίζε ανέφερε, παραμένουν κάποια ανοιχτά ζητήματα. Να διευκρινίσω λοιπόν ότι η θέση σε ισχύ του κανονισμού θα γίνει 20 ημέρες μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφόσον ψηφιστεί, όμως ε, η εφαρμογή του ξεκινάει τέσσερις μήνες μετά την θέση σε ισχύ του. Επομένως, αν όλα πάνε κατευχήν, ε, μπορούμε να αναμένουμε ότι θα αρχίσει να εφαρμόζεται την, άνοιξη του 2018, όχι λοιπόν 1η Ιανουαρίου του 2018. Έρχομαι τώρα στις συγκεκριμένες ανησυχίες που έχουν εκφραστεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται πριν την θέση σε εφαρμογή ε, αυτού του κανονισμού να δημοσιοποιήσει ξεκάθαρες ε, κατευθυντήριες οδηγίες που θα ξεκαθαρίζουν ακριβώς ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να λάβουν τι είδους μέτρα. Ε, ποια μέτρα. <clears throat> Επί τη ε, βάση των προβλέψεων του άρθρου 2 και της συζήτησης που έγινε στις 19 Ιουλίου στη Διαρκή Επιτροπή. Αυτό αναφέρεται επίσης ξεκάθαρα και στα πρακτικά της Επιτροπής. Μπορώ λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι θα είναι απολύτως ξεκάθαρες οι οδηγίες και θα είναι απολύτως ξεκάθαρες στις επιχειρήσεις ε, ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους. Όσον αφορά τη χρήση χρωματικών οδηγών. είναι ένα εύχριστο και απλό εργαλείο για να εξασφαλίσει κανείς ότι η ποσότητα ακριλαμιδίου σε ένα τρόφιμο είναι κάτω από τα όρια. Για παράδειγμα, σε ένα ξενοδοχείο το πρωί, στο, πρωινό, αν κάποιος ψήσει τη, τη, τη φέτα του τόστ υπερβολικά πολύ, δεν είναι δυνατόν να θεωρήσουμε ότι είναι υπεύθυνο ο ιδιοκτήτης του, ξενοδοχείου για αυτό το λάθος που κάνει ο πελάτης του. Άρα φυσικά, ε, εάν κάποιος ε, καταναλωτής αγνοήσει αυτό που του δείχνει ο χρωματικός οδηγός, ε, δεν θα ευθύνεται για αυτό ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Διευκρινίζεται επίσης ότι η ρηγματοληψία μπορεί να γίνεται κεντρικά, γιατί οι επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων έχουν τυποποιημένες διαδικασίες. Δεν χρειάζεται αυτή η δειγματοληψία. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα λόγος να γίνεται σε κάθε εστιατόριο, σε κάθε επιχείρηση του κλάδου της εστίασης σε ολόκληρη την Ένωση. Αυτή η δειγματοληψία και αυτή η ανάλυση μπορεί να γίνει με τρόπο αναλογικό. Θεωρούμε λοιπόν ότι το προσχέδιο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξασφαλίζει τη δημόσια υγεία, τηρώντας παράλληλα τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας. Έχει υποβληθεί ένα αίτημα να αναβληθεί η ψηφοφορία για η πρόεδρος παρεμβαίνει, δεν το ανέφερα αυτό Συγγνώμη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα αποφασίζουμε αν θα ψηφίσουμε ή όχι σήμερα. Αλλά πρώτα θα μιλήσουμε για τις προβλε... προβολές, για τις αντιρρήσεις μάλλον, για τις ιδιότητες ενδοκρινικών διαταρακτών. Και παρακαλώ, όποιος λάβει το λόγο, γιατί όλοι μας θα κερδίσουμε, να είναι όσο δυνατόν πιο σύντομη η κυρία Γκούντελαντ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και θα είμαι όσο δυνατόν σύντομα. Αντίρρηση λοιπόν έχω προς το σχέδιο πράξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Κανονισμό Φυτοπροστασίας που ορίζει κριτήρια για τον ορισμό των ιδιωτήτων ενδοκρινικής διατάραξης γιατί, και για να είμαι σαφής η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής βέβαια δεν δεν είναι ολόκληρη κακή αλλά δεν είναι και τόσο καλή και, τόσο, και πάνω απ' όλα δεν έχει υγεία νομική βάση. Η νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος έχει ανακαλύψει ότι έχει ξεπεράσει με την εισαγωγή από μιας νέας παρέκκλησης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εντολή τη για τους οργανισμούς αυτούς το 382 του δεύτερου παραρτήματος. Ο σχετικό κανονισμός αυτή τη στιγμή ορίζει ότι η ενεργό ουσία θα εγκρίνεται μόνο εφόσον αποδειχθεί, θεωρείται ότι δεν έχει ενδοκρινική ε, ιδιότητες ενδοκρινικής διατάραξης και δεν ε, παραβλάπτει τους ε, οργανισμούς στόχους με ρεαλιστικές συνθήκες χρήσεως πλην των περιπτώσεων που είναι πραγματικά μελιτέα η διατάραξη. Ε, η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως εισάγει μια παρέκκληση στο σημείο αυτό και αφήνει ανοιχτό ένα παραθυράκι. Με την αλλαγή ενό ουσιώδου στοιχείου του κανονισμού παραβιάζει σαφώ τις εξουσίες που τις έχουν εκχωρηθεί. Παράνομα. Και σε αυτό πρέπει να τη δράσουμε. Ιδιαίτερη σημασία βέβαια έχουν τα επιστημονικά στοιχεία για την ενδοκρινική διατάραξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα λέει ότι υπάρχει κίνδυνο περαιτέρω καθυστερήσεων αν δεν εγκριθούν τα κριτήρια και ότι ω εκ τούτου το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποδεχθεί την πρόταση. Εμεί θα πούμε όμω ότι. και πρέπει να το θυμόμαστε αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι η Επιτροπή όφιλε να έχει ήδη το Δεκέμβριο του 2013 καταθέσει τα σχετικά κριτήρια. Μην ξεχνάμε ότι η Επιτροπή μάλιστα έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διότι δεν ε, ήρθε στο ύψος των υποχρεώσεων της και δεν έκανε σωστά τη δουλειά της. Της καθυστερής λοιπόν δεν της έχει προξενεί στο Κοινοβούλιο. Του έχουμε επανειλημμένως καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση και τώρα έρχεται η Επιτροπή να καταθέσει κριτήρια τα οποία δεν ευθυγραμμίζονται με τα όσα ε, προβλέπεται στην ε, εντολή της Επιτροπής, με τόσα προβλέπονται στην εντολή της Επιτροπής. Έτσι λοιπόν, βεβαίω έχει καθήκον να μας προστατεύει από τις κίνδυνες ουσίες. Ο πολίτης Ευρώπης δεν ε, μπορεί να εκβιάζεται με αυτά τα διαδικαστικά εκβιαστικά διλήμματα. Το Κοινοβούλιο δεν θα πέσει στην παγίδα. Δεν θα δεχθεί κριτήρια μη εδρεωμένα επιστημονικά μόνο και μόνο επειδή η Επιτροπή καθυστέρησε τόσα χρόνια. Λοιπόν, ζητούμε νέα πρόταση, χωρίς παρεκκλήσεις, που δεν θα φέρει στα συνέπεια την ανάγκη η Επιτροπή κάθε πράγμα να το, να το επανεξετάσει, αλλά θα αποκαταστήσει την παρανομία παρατυπία. Παρακαλώ, κύριο Σεκάουτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι και εγώ σύντομο γιατί μπορεί να παρασυρθεί κανεί ε, και να αρχίσει να μιλάει για 7,5 χρόνια ε, τόσο, μεγάλο, τόσο πολύ έχουν κρατήσει αυτές τις συζητήσεις. Το θέμα εδώ είναι για όλους μας. Έχει υπερβεί το όρια της εντολής της Κομισιόν, ναι ή όχι. Είναι θέμα κράτους δικαίου όλο αυτό. Δεν έχει να κάνει με το περιεχόμενο. Ο καθένας μας έχει διαφορετικές πολιτικές απόψεις, τις γνωρίζουμε, αλλά το ερώτημα είναι η Κομισιόν έχει υπερβεί τις εξουσίες της. Γι' αυτό ζητάμε μια νομική γνωμοδότηση για το θέμα αυτό. Θα μας βοηθήσει να δούμε κατά πόσο συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η νομική γνωμοδότηση λοιπόν καταλήγει σε ένα πολύ σαφές συμπέρασμα ότι η Κομισιόν υπερβαίνει τις εξουσίες της. Τελεία και παύλα. Τώρα κάποιοι λένε ας είμαστε ρεαλιστές. Αλλά εδώ ξέρετε μιλάμε για κράτος δικαίου και όσοι υποστηρίζουν το κράτος δικαίου και το νόμο και την τάξη ε, και τώρα δεν του πειράζει που η Κομισιόν υπερβαίνει τι εξουσία τη. Αυτό δεν έχει νόημα και το θέμα είναι σε ποιο σημείο υπερβαίνουν. Στα κριτήρια αποκλεισμού. Τα κριτήρια αποκλεισμού ήταν το θέμα συζήτηση το 2009 όταν ο κανονισμό ε, τέθηκε επιτάπητος. Πώς θα ορίζονταν τα κριτήρια αποκλεισμού, δηλαδή υπήρχαν ε, ορισμοί για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και μετά τίθεται το ερώτημα του πότε θα εφαρμόζονται και εκεί ορίζονται τα κριτήρια αποκλεισμού. Γι' αυτό ε, καταρτίστηκε ένα ε, τεράστιο παράρτημα που ορίζει τα κριτήρια αποκλεισμού και τα, στο παράρτημα αυτό λέει σαφώς ότι θα εγκρίνεται μόνο εφόσον δεν έχει ενδοκρινικές διατρακτικές ιδιότητες σε ορισμένους οργανισμούς. Αυτή η διάταξη την αλλάζει τώρα η Κομισιόν, δημιουργώντα μια εξαίρεση από αυτέ. Όταν θέλει κανεί να κάνει μια εξαίρεση σε ένα ουσιώδε στοιχείο του κανονισμού, αυτό πρέπει να γίνει με συναπόφαση. Και η Κομισιόν τώρα λέει τα χρειαζόμαστε γρήγορα, μετά από 7,5 χρόνια τη ήρθε. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Δεν συζητάμε εδώ τα κριτήρια. Το κομμάτι αυτό της πρότασης το, στείλ, το στείλαμε. Αν θέλουμε εξαίρεση, πρέπει να μας κάνετε μια πρόταση που θα ψηφιστεί με συναπόφαση, που θα αποφασιστεί με συναπόφαση. Ε, και στην νομική γνωμοδότηση καθίσταται σαφέ ότι αυτά τα κριτήρια αποκλεισμού στο παράρτημα αποτελούν ουσιώδη στοιχείο του κανονισμού αυτού. Διότι καμιά φορά έρχεται η Επιτροπή και μα λέει Μα δεν είναι παραπαράρτημα αυτό που αλλάζουμε. Πρώτα απ' όλα είναι εξουσία της Κομισιόν. Μπορεί ξαφνικά να αποφασίσει η Κομισιόν η ίδια κατά πόσο ένα στοιχείο είναι ουσιώδες ή όχι. Και δεύτερον, ένα παράρτημα, όπως γνωρίζουμε πολλοί από εμά, μερικές φορές είναι στοιχείο κλειδί. Ένα ουσιώδε η οχι και δευτερον ενα παραρτημα οπως γνωριζουμε πολλοι απο εμα μερικε φορε στόχη για ε, ε, τι ανανεώσιμες πηγέ ενέργεια για το κάθε κράτος μέλος ε, στην οδηγία για τι ανανεώσιμες πηγέ ενέργεια. Δεν μπορεί να πει κανεί ότι αυτό δεν είναι ουσιώδε στοιχείο του κανονισμού, οπότε το επιχείρημα σε αυτό είναι αβάσιμο κομισιόν. Αν θέλετε να αλλάξετε, να κάνετε αλλαγή. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε. Θα τσακωθούμε για το περιεχόμενο, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με διαδικασία συναπόφασης και όχι με εκτελεστική πράξη. Αυτή είναι η βάση, αυτό είναι το θέμα. Οπότε παρακαλώ τους συναδέλφους να βάλουμε στην άκρη τις πολιτικές μας ιδεολογίες και να δούμε τη νομική πτυχή όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερβαίνει τις εκτελεστικές εξουσίες. Έχουμε και νομική γνωμοδότηση που το επικυρώνει και ζητώ συγγνώμη που τώρα 7,5 ε, ε, ε, χρόνια η Κομισιόν κινείται προς μια κατεύθυνση και τώρα την αλλάζουμε, αλλά επιμένω. Εάν το αφήσουμε θα κάνουν και άλλα και άλλες τέτοιες υπερβάσεις των εξουσιών τους. Οπότε ως Κοινοβούλιο πρέπει εδώ να τραβήξουμε μια νομική κόκκινη γραμμή. Εγώ σας τραβάω μια χρονική γραμμή αυτή τη στιγμή. Σας παρακαλώ συνάδελφοι. Τηρείτε το χρόνο σας. Κύριε Αντελάη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η πρόταση που έχουμε μπροστά μας σίγουρα δεν είναι τέλεια. Ωστόσο αξίζει να υπάρχει. Μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε ε, με, μια, με την αυστηρότερη νομοθεσία στον κόσμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ορισμοί είναι ορισμοί ε, που έχουν επικυρωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Τι ζητάμε παραπάνω. Τώρα, ας είμαστε ρεαλιστές, πρέπει να είναι δυνατή η εφαρμογή των ορισμών αυτών στις, ε, στα νομικά μας συστήματα και τώρα ε, έχει περάσει πολλής χρόνος πια, πρέπει να προχωρήσουμε. Ζητάμε αυτούς τους ορισμούς εδώ και πολύ καιρό είναι απαραίτητη και του χρειαζόμαστε σήμερα. Αν ε, πετάξουμε στα σκουπίδια αυτή την πρόταση, ξεκινάμε για άλλη μια δεκαετία διαπραγματεύσεων. Όταν λέμε θέλουμε έναν ορισμό, είναι σημαντικό και αναγκαίο για την προστασία των πολιτών, τότε σα παρακαλώ, σα συγκετεύω, μην ε, ανοίγουμε μια συζήτηση που θα διαρκέσει άλλη μια δεκαετία. Δεν είναι τέλεια τα πράγματα, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να προχωράμε, Προστατεύοντα την υγεία, ε, ενθαρρύνοντα την καινοτομία για όλα αυτά χρειάζονται αυστηροί και σαφείς κανόνες. Οι παραγωγοί βιομηχανοί πρέπει να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, πώς θα ε, παράγουν προϊόντα πιο ασφαλή για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ που τηρήσατε το χρόνο, κυρία Γκέρλινγκ. Κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ. έχω ετοιμάσει ένα μακροσκελή λόγο αλλά θα δείξω αυτοσυγκράτηση. Θέλω να πω ότι δεν υποστηρίζω το την ε, πρόταση ψηφίσματος, λέει ο Μιλήτρια. Θεωρούμε ότι είναι αποδεκτή και τη μη τέλεια η πρόταση της Επιτροπής. Όπως είπε είναι κάτι το οποίο επί χρόνια μας απασχολεί. Πρέπει πια να να καταλήξουμε με βάση αυτά που έχουμε στο τραπέζι και να μην ψάχνουμε λόγους να, το, να καθυστερήσουμε περισσότερο την υπόθεση, ε, μπορεί να έχουν μόνο σε οργανισμούς στόχους ε, συνέπειες αυτοί οι διαταράκτες, παραδείγματι σε ασθένειες ε, των φυτών, οπότε μπορούν να χρησιμοποιούνται ακόμη. Ταυτόχρονα, εάν δεν ε, έχουν κατανεμηθεί ως, δεν έχουν καταχωριστεί ως διαταράκτες οι ουσίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα. Μάλλον δεν έχουν καταχωριστεί ως, ως ε, ασφαλείς. Δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι διαταράκτες και έτσι δεν μπορούμε να είμαστε τόσο απόλυτοι. Η ε, αντικατάσταση του κριτηρίου παράβλαψης ε, πρέπει να γίνει. Ιδάλλως θα παραμένει η αβεβαιότητα για πολύ καιρό, θα καταχωρούνται σε λάθος σημείο, ε, θα καταχωρίζονται σε λάθος σημείο ουσίες. Και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε και να φέρουμε αποτελέσματα. Για δε την ε, γνωμική πραγματογνωμοσύνη που μας ανέφερε ο Μπάρς. Ναι, σημαντικό είναι και το κράτος δικαίου βέβαια, αλλά Σα είπα ότι πρόκειται για πραγματογνωμοσύνη. Άρα είναι μόνο μία γνώμη και τίποτα παραπάνω. Νόμο δεν είναι σίγουρα. Ευχαριστώ, κύριε Ρή. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Βέβαια, ξέρετε, έγινε λόγος για γενετικά τροποποιημένους οργανισμός για γλυφοζάτη. Τώρα είμαστε στους ενδοκρινικούς διαταράκτες, δηλαδή είμαστε στο κέντρο των ανησυχιών των Ευρωπαίων πολιτών. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η συζήτηση. Δυστυχώς ε, είναι στην καθημερινή μας ζωή παρόντα αυτά τα στοιχεία. 800 ε, προϊόντα, χημικές ουσίες έχουν καταγραφεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας πως μπορεί να επηρεάζουν το ορμονικό μας σύστημα. Έτσι λοιπόν είναι και ήταν πάντοτε πολύ σημαντική η διαμόρφωση ενός νομικού πλαισίου μετά τη συμφωνία της 4ης Ιουλίου, αν δεν απατώμε, για τα χημικά, που μετά από πολλές καθυστερήσεις, αναβολές και άλλες δυσκολίες μπόρεσε να καταλήξει σε μια έννοια νομικού προσδιορισμού που θα έπρεπε κανονικά να μας εξασφαλίζει ασφάλεια δικαίου, αλλά δεν τα καταφέρνει γιατί η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου μας λέει ότι είναι σαφής η υπέρβαση των καθηκόντων και εξουσιών από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα επαναλάβω τα ε, σχόλια και την αιτιολόγηση όλης αυτής της υπόθεσης που μας εξέθεσαν οι συντάκτες και ο Μπάρς, αλλά πάντως εδώ έχουμε να κάνουμε μια αντιπαράθεση νομικού ε, χαρακτήρα μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου είναι σαφές πως ε, δεν υπάρχει καμία πρόθεση για ένα φιλόδοξο έργο ε, με όλες αυτές τις παρεκκλήσεις που αφορούν ακόμη και ζυζανιοκτόνο που μπορεί να έχει ε, πολλαπλές ενδοκρινικές διαταράξεις ως συνέπεια στον οργανισμό των εντόμων έχουμε να κάνουμε με σοβαρά σοβαρή αμέλεια. Έτσι λοιπόν χρειάζεται μια στρατηγική για όλους αυτούς τους διαταράκτες που βρίσκονται παρόντες παντού στη συσκευασία, τα πλακτιστικά, τα παιχνίδια, παρόντες παντού στην καθημερινή μας ζωή και πρέπει να εξασφαλιστεί μια νομοθεσία όπως είδατε. Ήμουνα σύντομη γιατί μίλησα τόσο γρήγορα και νομίζω ότι πρέπει να υπερψηφίσουμε αυτήν την αντίρρηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χάζενκαμπ. Ε, dank u wel, σας ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζουμε ότι αυτοί ε, οι ενδοκρινικοί διαταράκτες αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη. Και για το αναπαραγωγικό σύστημα και μερικές φορές οδηγούν και σε καρκίνο. Επομένως, πρέπει να ε, τους περιορίσουμε, να, να αναλάβουμε δράση επί τη βάση κριτηρίων. Δυστυχώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλήγει σε ένα κατάλογο κριτηρίων που ε, έχει καθυστερήσει, δεν βρίσκοντας την αρχική πρόταση. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν υποστηρίζουμε τι αντιρρήσει. Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα εδώ. Πρώτα απ' όλα, ποιος φέρει το βάρος της απόδειξης. Ε, το βάρος της απόδειξης είναι ξεκάθαρο για τις περιπτώσεις των και ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία υφίσταται ήδη δεδομένου, δεδομένου ότι αυτά τα προϊόντα βρίσκονται ε, ήδη στην ε, αγορά. Για άλλα είδη προϊόντων, όπως για παράδειγμα για τα παιχνίδια ή για τους τεχνητούς χλωτάπητες που είναι χρησιμοποιούνται σε παιδικές χάρες, όπου χρησιμοποιούνται μια σειρά από φαινόλες που πιθανώς να είναι επικίνδυνες και εδώ πρέπει να αναλάβουμε δράση για τον περιορισμό αυτών των ουσιών. Αναλύεται μια λίστα κριτηρίων, μήπως θα ήταν πολύ πιο απλό να απαγορεύσουμε τη χρήση όλων αυτών των προϊόντων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι προφανές για μας ότι η Επιτροπή υπέκυψε στις πιέσεις των μεγάλων επιχειρήσεων της χημικής βιομηχανίας και της ιουργικής βιομηχανίας. Ε, ωστόσο υπάρχουν ε, επιστημονικά κριτήρια για τους, επιστημ... για ενδοκρινικούς διαταράκτες και αυτά πρέπει μόνο με αντικειμενικό τρόπο να αξιοποιηθούν με βάση λέει, τα στοιχεία που αναφέρονται στο ενδοκρινικό σύστημα και ανεξαρτησία οδήποτε άλλο μελήματος και δι Αν κοιτάξουμε λοιπόν το κείμενο που έχει υιοθετηθεί, εξετάζονται και θεωρούνται ενδοκρινικοί διαταράκτες μόνο εκείνες οι ουσίες για τις οποίες έχει αποδειχθεί σχέση αιτίας και αίτημα του μεταξύ της ουσίας και της ζημιάς στον οργανισμό. Δηλαδή δεν λαμβάνεται καμία πρόνοια για τις ουσίες για τις οποίες υπάρχει ε, υποψία ε, ζημιογόνου δράση στον ανθρώπινο οργανισμό. Παραβιάζει ω εκ τούτου την αρχή τη πρόληψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό παράπτωμα και γι' αυτό αντιτίθεμαι στην πρότασή τη. Κύριο Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε συστήσει πολλές φορές το θέμα των ενδοκρινικών διαταρακτών οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις αλλά και η βιομηχανία δεν είναι ικανοποιημένες με την πρόταση της Επιτροπής. Είναι μια συμβαστική πρόταση στην οποία έχουν συμφωνήσει τα κράτη-μέλη όσον αφορά όμως μόνο την έκτακτη διαδικασία. Μπορούμε να συζητούμε και να διαφωνούμε για τα νομικά ζητήματα, ωστόσο πρόκειται για ένα δημόσιο διάλογο, ο οποίο έχει κρατήσει χρόνια, έχουν εκφραστεί 30.000 αντιρρήσεις, έχει κρατήσει χρόνο, έχει κοστίσει χρήμα και καλείται τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ταχύτερο δυνατό να διατυπώσει νέα πρόταση. Μα είμαστε και σοβαροί. Όποιο το ζητάει αυτό ξέρει πολύ καλά ότι θα κρατήσει χρόνια υπόθεση, 4-5 χρόνια. Δηλαδή θα έχει ξεπεράσει και τη δική μα τη βουλευτική εντολή. Ε, δεν είναι αυτό ο καλύτερο τρόπο να ε, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Συγκρίνουμε αυτό το οποίο βρίσκεται ε, ω πρόταση στο τραπέζι για να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου για τη βιομηχανία και η προστασία των πολιτών. Δεν υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι, άλλωστε και οι πράσινοι ε, έχουν υποβάλει στην ε, Γερμανία, στη γερμανική κυβέρνηση αντίστοιχη επίκαιρη ερώτηση, ίσως, ε, την οποία δεν μπορώ τώρα να σας εκθέσω διότι δεν έχουμε το χρόνο, αλλά ο φίλος Μπάρτας ρωτήσει τους Γερμανούς συναδέλφους του και πολιτικού του φίλου θα του πούνε. Άλλωστε, μέσα από την συνεργασία τώρα για το συνασπισμό Τζαμάικα, τον τρικομματικό στη Γερμανία, νομίζω ότι θα αμβληθούν όλε του οι αντιρρήσει. Η κυρία Γκροστέτ. Κοίταξε, το θέμα εδώ είναι να προστατεύσουμε την ε, υγεία των συμπολιτών μα. Όλοι εδώ και χρόνια ε, επιμένουμε να λυθεί κάποια θέση για του ενδοκρινικού διατράκτε. Και τώρα πλέον έχουμε μια θέση, σίγουρα δεν είναι απόλυτα ικανοποιητική. Μακράν εγώ θα προτιμούσα την πρόταση με τα ζυζανιοκτώνα και να υπάρχει μια εξαίρεση για τα προϊόντα που μπορούν να θεωρηθούν ε, που ε, ε, έχουν αποτέλεσμα ενδοκρινικού διαταράκτη, αλλά τα πράγματα δεν είναι άσχημα. Έχουμε μια πρόταση. Ήδη είναι ένα σημαντικό βήμα γιατί περιμένουμε εδώ και χρόνια και τώρα ε, μπορούμε να πούμε τα απορρίπτουμε όλα αυτά, θέλουμε περισσότερα. Ναι, ενδοκρινικοί διαταράκτες, όλοι θέλουμε να κάνουμε περισσότερα για αυτούς. Αλλά εδώ έχουμε κάνει ένα πρώτο βήμα, το οποίο είναι ένα, κάτι σημαντικό. Μπορούμε να συνεχίσουμε ε, να ασχολούμαστε με το ζήτημα, αλλά το να απορρίψουμε αυτή την αντίρρηση θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Είμαι υπέρ της πρότασης της Κομισιόν. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν τόσο σύντομοι. Ο κύριος Μπέρεντ από την Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι σύντομος όπως και οι υπόλοιποι. Θα μπορούσα να πω πολλά για την επιχειρηματολογία που ακούσαμε ε, στο σχέδιο αντίρρησης, αλλά θα επικεντρωθώ κυρίως σε αυτή την ρήτρα ε, εξαίρεσης, όπως ονομάστηκε, στο derogation clause που φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο του θέματος. Να σας υπενθυμίσω όμως πρώτα ότι πράγματι η διαδικασία υπήρξε μακροχρόνια και περίπλοκη. Ε, το να υποβάλει αυτά το σχέδιο κριτηρίων ε, η Κομισιόν ε, και εδώ τώρα στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο για αναθεώρηση. Ξέρετε, υπάρχουν πολλέ και διαφορετικέ απόψει για το θέμα αυτό. Οπότε αυτό που προτείνουμε είναι η καλύτερη συμβαστική που μπορούσαμε να σχεδιάσουμε. Τώρα για αυτό το συγκεκριμένο σημείο, ότι η ρήτρα αυτή που βρίσκεται στο επίκεντρο τη αντίρρηση, πρέπει να υπογραμμίσω ότι αντίθετα με την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου, η νομική υπηρεσία τη Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα Σαφώ ότι έχουμε τέτοια εξουσία και ότι το σημείο στο 382 δεν είναι ουσιώδη στοιχείο, αντίθετα με τα άλλα κριτήρια αποκλεισμού που αναφέρονται σε ένα άρθρο του κανονισμού. Αυτό δεν είναι ουσιώδη στοιχείο. Δεν υπάρχει τίποτα στα άρθρα ή στι ιτεολογικέ σκέψει που να περιορίζει το Κοινοβούλιο ή την Κομισιόν ε, όσον αφορά τα άλλα σημεία του παρατήματος Γι' αυτό το νομικό επιχείρημα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο κανονισμός γενικότερα έχει το στόχο να προωθήσει την ανάπτυξη και την θέση στην αγορά ουσιών που είναι πιο καλές από άλλες για την υγεία. Και οι Instant Growth Regulators θεωρούνται καλύτεροι, όπως καλύπτω από αυτή την ρήτρα και ε, είναι ουσιώδη στοιχείο στο IPM και υπάρχουν συγκεκριμένε απαιτήσει ε, δεδομένων ώστε να επιτρέπεται η ανάπτυξή του. Οπότε με το να του απαγορεύσουμε απλά χωρί καμία δυνατότητα εξαίρεση, ουσιαστικά δράμε κατά των στόχων ε, του κανονισμού στο σύνολό του. Τέλο θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι αυτή η συγκεκριμένη ρήτρα ήταν απολύτω απαραίτητη ώστε να επιτευχθεί η υποστήριξη ειδική πλειοψηφία στη Μόνιμη Επιτροπή. Ο κ. Σαϊκόλτ είπε ότι το χρησιμοποιώ ως απειλή. Δεν είναι απειλή, είναι γεγονός. Χωρίς αυτή τη συγκεκριμένη ρήτρα δεν θα είχαμε επιτύχει την ειδική πλειοψηφία στη Μόνιμη Επιτροπή και αντίθετα από ό,τι μας προτείνει η αντίρρηση δεν μπορούμε να επανέλθουμε με το ίδιο κείμενο χωρίς αυτή τη ρήτρα διότι δεν πρόκειται κάτι τέτοιο να λάβει την απαραίτητη υποστήριξη όπως είπαν και άλλοι ομιλητές, θα κολλήσουμε με τα ενδιάμεσα κριτήρια για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αν υπάρχει μία συνένεση σε αυτή τη συζήτηση, είναι αυτή. Τα ενδιάμεσα κριτήρια δεν είναι κατάλληλα για τον σκοπό. Καθορίζουν, ε, ε, εντοπίζουν λάθος στοιχεία, ε, λάθος ουσίες και όχι αυτές που είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες. Για να συνοψίσω, ενώ λοιπόν η πρόταση για τα μαθιά πολλών δεν είναι τέλεια ή αποτελεί σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Αυτό αποτελούν αυτά τα κριτήρια. Ένα σημαντικό βήμα προ τα μπρος με τα ενδιάμεσα κριτήρια. Και έχουμε προτείνει και μια ρήτρα αναθεώρηση ε, ε, μετά από την εμπειρία που θα έχουμε με την εφαρμογή αυτών των κριτηρίων. Οπότε μπορούμε να τα αναπτύξουμε περαιτέρω και να τα αναθεωρήσουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much. That... Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ ολοκληρώνω τη συζήτηση για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Πάμε στην ψηφοφορία. Πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία, έχουμε προβλέψει κάποια αρχαία για την ψηφοφορία σήμερα αλλά έχουμε λάβει δύο αιτήματα για, τη, για αναβολή της ψηφοφορίας ε, οπότε πρέπει να υποβάλω αυτά τα αιτήματα σε εσά. Το πρώτο αίτημα αφορά την αναβολή της ψηφοφορίας για το ακριλαμίδιο και όπως κατάλαβα από τη συζήτηση υπάρχουν αντιρρήσεις για την αναβολή της ψηφοφορίας, οπότε πρέπει να ψηφίσουμε επί του αιτήματος αναβολής. Ποιος είναι υπέρ του να δεχθούμε την πρόταση αναβολής της ψηφοφορίας για το ακριλαμίδιο στις 12 ε, Οκτωβρίου. Ας το κάνουμε ηλεκτρονικά. Είναι ευκολότερη η καταμέτρηση. Είναι η πρώτη ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Does everyone uh, have its card and voted? Έχουν ψηφίσει άπαντες. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Οπότε θα το ψηφίσουμε σήμερα. Η δεύτερη πρόταση που λάβαμε για αναβολή αφορά την ε, διεθνή ε, διακυβέρνηση των ωκεανών και αναβολή της ψηφοφορίας. Υπάρχουν αντιρρήσεις όσον αφορά την αναβολή αυτής της ε, ψηφοφορίας. Το αίτημα έγινε από τον εισηγητή. Δεν βλέπω να υπάρχει αντίρρηση, οπότε θα εγκρίνουμε αυτή την πρόταση. Οπότε η ψηφοφορία για τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών θα αναβληθεί έω την συνάντηση του Νοεμβρίου. Ξεκινάμε λοιπόν τι ψηφοφορίες. Το πρώτο στοιχείο είναι μια ψηφοφορία. Είναι η ψηφοφορία για την ε, γενετικά τροποποιημένη σόγια FG72 και τα λοιπά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. And the vote is closed. συγκρίνεται. Δεύτερο θέμα. Αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί για, τη γενετικά για την οτικά τροποποιημένους φασίλους φιόγιας. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τρίτη ψηφοφορία για σήμερα. Αντιρρήσεις. Σε σχέση με τα μέτρα περιορισμού και τα κατόφλια για με, στόχο την μείωση του ποσοστού ακριλαμιδίου στα τρόφιμα. Έρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Επόμενη ψηφοφορία. Αντιρρήσεις για τα κριτήρια σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Ψηφίστε παρακαλώ. the ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Επόμενη ψηφοφορία. για τον κανονισμό μέσω του οποίου εγκρίνονται νομικές πράξεις σχετικά με το άρθρο 2, τη βάση του άρθρου 291 της συνθήκης. Πρώτα θα ψηφίσουμε τις α, τροπολογίες ομού, 1 έως 3, υπέρ, κατά, εγκρίνονται. Τροπολογίες 1 έως 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 1.26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 129 και 130 καταπίπτουν, ναι, ωραία. Μια ναι, ε, 195 υπέρ. Ε, 159, συγγνώμη. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 124 και 127 Τα αποχές, απορρίπτονται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική. Ψηφίστε παρακαλώ. Εγκρίνεται. Τώρα θα πρέπει να ψηφίσουμε ε, επί της επιστολής που θα στείλω ως πρόεδρος της Επιτροπής μας, ε, στην οποία θα επισυνάψω ε, την τροπολογία την οποία μόλις υπερψηφίσαμε. Ποιος είναι υπέρ αυτής της επιστολής, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. There is one more. Let me find it. We vote on implementation of e Ψηφοφορία για την εφαρμογή της μακροπεριφερειακής στρατηγικής. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές. σε ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίστε για την τροπολογία 9 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά εποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Εποχέ. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Εποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Εποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Εποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά απο, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβεβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30, ε, ε, συγγνώμη, 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 Αποχέ. Α ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε για την τροπολογία 47 παρακαλώ. The vote is closed. Πέρασε εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 50 υπέρ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 while uh, you will uh, stay with us or leave, but nevertheless try to... Άντε να δούμε ποιος θα μείνει κοντά μας σήμερα. Όσοι θέλετε παρακαλούμε, ή λυπή, κατεβάστε λίγο την ένταση για να συνεχίσουμε. Colleagues and the other participants at this meeting, would you please... Οι συνάδελφοι και οι λοιποί. Παριστάμενοι παρακαλούμε. Και ευχαριστούμε. Ανακοινώσεις λοιπόν, διάφορα θέματα. Πρώτα απ' όλα, έχει εντοπιστεί σφάλμα σε κανονισμό για τη διάθεση στην αγορά και χρήση βιοκτώνων αφορά την ενεργό ουσία του παραρτήματος 1 ε, κατηγορίας 6, τρίτη γραμμή του πίνακα και τα σχετικά παραπεμπτικά νούμερα. Το Κοινοβούλιο κλήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίε του Συμβουλίου να συμφωνήσει στην προτινόμενη διόρθωση του σφάλματος αυτού. Έτσι λοιπόν, έχει ετοιμαστεί κείμενο παροραμάτων για το κείμενο, για το πίνακα. Προβλέπεται από τον κανονισμό. Απεστάλλει το κείμενο των παροραμάτων την Τετάρτη σε όλους τους ενδιαφερομένους και αν δεν εκφραστούν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος συνεδρίασης θα θεωρηθεί πως εγκρίνεται η διόρθωση και θα, ενστομα... και θα προβλεφθεί για ανακοίνωση στην ε, πρώτη ολομέλεια του Οκτωβρίου. Άλλο θέμα. Σύνθεση της ε, ομάδας διαπραγμάτευσης Λουλουσιεφ. Κατόπιν της αποφάσεως της Ολομέλειας για την αναπομπή του φακέλου Λουλουσιεφ με βάση το άρθρο 69 σίγμα τάφο της ομάδας προεδρεύει η πρόεδρος με συμμετοχή εισηγητού και σκιωδών. Τρίτον, ETS αεροπορία. Κατόπιν αποφάσεω τη Ολομελία να αναπέμψει στην Επιτροπή Περιβάλλοντο για την ανάληψη διαπραγματεύσεων του ε, τη προτάσεω για τι ανταλλαγέ ε, εκπομπών στην αεροπορία. Ορίζεται ομάδα προεδρευομένη από τον πρόεδρο με μέλη των εισηγητή και του σκιώδη εισηγητέ συνεδριάσεις της ΕΝΒΗ, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Κατόπιν αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως για μια δοκιμαστική φάση κατά την οποία συνεδριάσεις τρίτες και τετάρτες στις ομάδες επιτροπών θα ξεκινούν στις 2 και 30, 2 και 30, 14 και 30, οι απογευματινές συνεδριάσεις στις 11 Οκτωβρίου Τρίτη, 21 Νοεμβρίου Τρίτη και 28 Νοεμβρίου Τρίτη. Οι απογευματινές συνεδριάσεις της Επιτροπής μας θα ξεκινήσουν στις 2.30 αντί για τις 3. 12 Οκτωβρίου, το απόγευμα, αποδεσμεύεται ο προγραμματισμός των ατουσών και συνεδριάσεων από την ε, προβλεφθήσα δοκιμαστικά συνεδρίαση. Εργαστήριο με τίτλο «Κύκλος ζωής των φυτών 2020» τον Οκτώβριο 10 με 12.30 όπως έχει σχεδιαστεί ενημερωτικά για τα μέλη της Επιτροπής μας ως προς την εφαρμογή του προγράμματος LIFE, πρώτα αποτελέσματα των ενοποιημένων έργων του προγράμματος LIFE. Παρακαλείστε όλοι να είστε παρόντες. Επίσης πρέπει να σας ενημερώσω για συνεχιζόμενες ε, θεσμικές δύο οργανικές ε, διαπραγματεύσεις και συνομιλίες. Πακέτο για την κυκλική οικονομία πρώτος, άτυπος τριμερής διάλογος για τα απόβλητα, ανταλλαγή απόψεων και διαπραγμάτευση έγινε για διάφορα θέματα. Ελήφθη απόφαση σε τεχνικό επίπεδο να παραπεμφθούν τα θέματα και ε, των αποβλήτων συσκευασίας και της ε, οδηγίας για τις χωματερές. Κάποια ζητήματα θα πρέπει να ξανασυζητηθούν σε πολιτικό αλλά και σε τεχνικό επίπεδο. Οι συμβιβασμοί, οι συμβαστικές λύσεις, οι οποίες, οι οποίες εξασφαλίστηκαν, ε, αποκλειωμένων των στόχων περιορισμού των, ε, της μείωσης των αποβλήτων, ε, παράρτημα 4α και επικίνδυνα απόβλητα αναβλήθηκαν οι κατανομές αναπροϊόν και απόβλητο και απόρριμα. Αυτά για την ε, δέσμη για τα απόβλητα. Οι διαπραγματεύσει για την οδηγία για τον περιορισμό των εκπομπών, ETS, Τέταρτος τριμερής διάλογος, τέταρτη φάση, περιορισμός των εκπομπών, 13 ε, Σεπτεμβρίου στο Κοινοβούλιο. Έτσι δεν είναι. Εξετάσαμε με βάση την εντολή της ε, Κορεπέρου 8 Σεπτεμβρίου τις κύριες δίκημες. Α, ναι, Στρασβούργο ήταν, ναι, ναι, ναι, γι' αυτό δεν προέδρευσαμε στο Κοινοβούλιο. Σημαντική πρόοδος ως προς τις διατάξεις ΕΝΕΣΑ προβάλλονται οι δικές μας προτάσεις για τη δοκιμαστική φάση περιορισμού των αδειών MSR στο Συμβούλιο. Καλώς ορίζουμε την πρόταση που ακούστηκε κατά τον τριμερή διάλογο, εντατικές συζητήσεις για το Ταμείο Καινοτομίας. Μάλλον έχουν εξασφαλιστεί κάποιες προσεγγίσεις θέσης των θεσμικών οργάνων. Σύμφωνα με σε διάφορα στοιχεία και δει εθελοντική κατάργηση σε περίπτωση κλεισίματος μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, επέκταση του καταλόγου διαρροής άνθρακα κλπ. Προσεχή στριμμένης διάλογος 12 Οκτωβρίου. ETS για την αεροπορία. Πρώτος τριμερής διάλογος, άτυπος, με πρώτη την παρουσίαση του σκεπτικού των θέσεων Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Η Προεδρία υπέγραψε την ανάγκη για ασφαλή δικαίου για τους εμπλεκόμενους φορείς, υιοθετώντας τις προτάσεις της Επιτροπής, κάθε αλλαγή θεωρείται δηλαδή πρόορη. Η Επιτροπή υποστήριξε τη διαδικασία δηλώνοντας τη βούληση να εξετάσει περαιτέρω βήματα ώστε να ε, προσεγγίσουν οι θέσεις των ε, εμπλεκομένων πλευρών. Περαιτέρω συζητήσεις ενδεχόμενη συμφωνία 18 Οκτωβρίου. Αυτά ήταν τα όλιγα λόγια για τους τριμερείς ε, διαλόγους που διεξήχθησαν πρόσφατα. Και τώρα πάμε στη συζήτηση και την ημερήσια διάταξη που προβλέπει να το βρω. Επαναδιατύπωση εσωτερική αγοράς ηλεκτρικών ειδών ή ηλεκτρική ενέργεια. μάλλον με τον κύριο Μπέλετ. Σχέδιο γνωμοδότηση και έχετε το λόγο. very much, uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εδώ ασχολούμαστε με τον κανονισμό και όχι με την οδηγία για την οποία είναι ο συνάδελφος Πότσος ε, αρμόδιος ε, και φυσικά αποτελεί όλο αυτό κομμάτι του δέσμης μέτρων για την καθαρή ενέργεια. Ε, επιτροπή της ουσίας είναι η ΙΤΡΕ όπως γνωρίζουμε αλλά ε, έτσι όπως έχει σχεδιαστεί και οργανωθεί η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας επηρεάζει και τους κλιματικούς στόχους οπότε η εμπλοκή της Επιτροπής μας είναι σημαντική. Τι αφορά το, η έκθεση αυτή η αναδιατύπωση αυτή, την ε, υιοθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη δυνατότητα ε, παροχής ε, της απαλλαγής της ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανθρακούς εκπομπές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και διευκόλυνση της ροής της ηλεκτρικής ενέργειας από τα μέρη που παράγεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο ως προς το κόστος. Ήθελα να πω κάτι για την εφεδρική δυνατότητα που θα απαιτηθεί, αλλά θα Επανέλθουμε σε αυτό αργότερα. Δύο-τρία σημεία προτείνουμε εδώ ε, που έχουν προτεραιότητα διότι όλες οι τεχνολογίες, οι ανανεώσιμες τεχνολογίες έχουν οριμάσει πλέον ε, και οριμάζουν όλο και περισσότερο και μπορούν να ε, υλοποιηθούν χωρίς επιδοτήσεις, χωρίς κρατική υποστήριξη, οπότε μπορεί να είναι λίγο πρόωρο για να αποφευχθούν ε, στρέβλωση Να, να, ε, θεωρήσουμε ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί αυτή η πολιτική. Οπότε στην τροπολογία 20 προτείνουμε προσεκτική ε, αξιολόγηση πριν αφαιρεθεί αυτή η πρόβλεψη προτεραιότητας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το άλλο που είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία αυτής της αναδιατύπωσης είναι το ζήτημα της επάρκειας των πορών και των μηχανισμών δυναμικότητας. Φυσικά όλοι είμαστε υπέρ της προσέγγισης της Κομισιόν. Θέλουμε να υπάρχει μια συντονισμένη ευρωπαϊκή μεθοδολογία. Αυτό αποτελεί ένα θετικό βήμα. Ωστόσο απαιτείται καλύτερη ενδεχομένω ισορροπία μεταξύ ευρωπαϊκής μεθοδολογίας και ε, ε, τοπικών ή εθνικών ιδιαιτεροτήτων. Προτείνουμε λοιπόν η αξιολόγηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο να συμπληρώνεται στο μέλλον με αξιολογήσεις πιο εστιασμένες ε, και επίσης εστιασμένες σε εθνικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες. Επιπλέον το θέμα της δυναμικότητας, του μηχανισμού δυναμικότητας θα διασφαλίσει την ασφάλεια εφοδιασμού. Είμαστε υπεπισμένοι ότι αυτοί οι μηχανισμοί δυνατότητας δεν μπορούν να αποκλειστούν. Θα πρέπει να εξετάσουμε φυσικά το κόστος για τους καταναλωτές. η εισαγωγή αυτών των μηχανισμών ε, δυναμικότητα θα πρέπει να βασιστεί σε συγκεκριμένου λόγου και φυσικά να ληφθεί υπόψη και το κόστο ε, όπω θα μεταφραστεί, όπως θα εμφανιστεί στου λογαριασμού των καταναλωτών. Όλα αυτά πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά. Ένα άλλο στοιχείο εδώ είναι ότι οι μηχανισμοί δυναμικότητα θα πρέπει να βασίζονται σε διαφανή κριτήρια ε, και με επαρκή ευελιξία. χωρί να αντίκυνται στου κλιματικού και ενεργειακού στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέψτε μου, κυρία Πρόεδρε, να αναφερθώ στα συγκεκριμένα, στο συγκεκριμένο κριτήριο, το οποίο είναι κάπω ευαίσθητο των 550 γραμμαρίων ε, διοξιδίου του άνθρακα ανά κιλοβατόρα ως πρότυπο ε, επιδόσεων ε, εκπομπών. Πρέπει να δούμε και τον τρόπο με τον οποίο ορίζεται αυτό το κριτήριο, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι οι στρόβιλοι ε, ανοιχτού κύκλου ε, έχουν εφεδρική δυναμικότητα, αλλά δεν ε, ανταποκρίνεται σε αυτό το κριτήριο άμεσα των 550 γραμμαρίων. Οπότε πρέπει να λάβουμε υπόψη το ρόλο αυτού του ανοιχτού, ε, ε της ανοιχτής διαμόρφωσης ε, και να χρησιμοποιήσουμε κάποια ευελιξία. Ε, στον καθορισμό αυτών των κριτηρίων. Το τελευταίο που ήθελα να αναφέρω δεν σχετίζεται άμεσα με την ΕΜΒΗ, ε, αλλά έμεσα. Είναι περισσότερο ε, θέμα που αφορά την Ήτρε. Είναι η TSO, οι φορείς μετάδοσης και τα επωνομαζόμενα περιφερειακά λειτουργικά κέντρα. Εμείς υποστηρίζουμε τον αποτελεσματικό συντονισμό των ευρωπαϊκών συστημάτων και θέλουμε να γίνουν βήματα για ε, συντονισμό των περιφερειακών αυτών κέντρων. Το θεωρούμε απαραίτητα, αλλά το θέμα που θέλουμε να θέσουμε και που έχουμε θέσει σε πολλές ε, τροπολογίες είναι κατά πόσο γίνεται αυτό ε, από πάνω προς τα κάτω. Εμείς προτείνουμε την αντίστροφη διαδικασία από κάτω προς τα πάνω. Αλλά Θα εκπονήσουμε δηλαδή αυτή την ιδέα της ευρωπαϊκής ε, ε, διαχείρισης της μεταφοράς από κάτω προς τα πάνω. Προσπαθώ να προβούμε σε διαρθρωτικές αλλαγές μέσω αυτών των περιφερειακών κέντρων δηλαδή. Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί στόχοι. Έχουμε υποβάλει πολλές τροπολογίες και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τις όποιες προτάσεις των συναδέλφων η προθεσμοί για τις τροπολογίες ε, θα, θα να αναφέρετε εσείς κυρία Πρόεδρε. Ε, αναμένω να ακούσω τις απόψεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπαλότ. Πάμε στους σκιώδεις εισηγητές. Ε, ο πρώτος είναι ο κύριος Πότσο. ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για αυτό το σχέδιο εκθέση. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Στην αρχή δεν μας έδωσαν καθόλου αυτό το θέμα και μετά βρεθήκαμε στη δύσκολη θέση να υπάρχουν δύο εισηγητέ ε, ουσιαστικά για το ίδιο θέμα. Ε, χαίρομαι λοιπόν που το σκεπτικό σας έμοιαζε με το δικό μου ε, στη δική μου έκθεση για την οδηγία. Συμφωνώ που ασχολείστε με τα περιφερειακά ε, κέντρα όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων. Αυτό αντιστοιχεί πράγματι στι αρμοδιότητες τους. Είναι σημαντικό αυτό. Από αυτή την άποψη η αλλαγή στα άρθρα αυτά θα πρέπει να ε, υπάρχουν και στο άρθρο 5 που αφορούν τη δυναμικότητα και τις προμήθειες. Θα πρέπει να μπορούν να παρέχουν ε, τοπικά. Οι TSO θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να παρέχουν εγχώρια ε, ηλεκτρική ενέργεια, αν αυτό είναι πιο αποτελεσματικό ως προς το κόστος και πιο ασφαλές. Ε, επίσης, καλό θα ήταν να αναλύσουμε κατά πόσο είναι αναγκαίο να υπάρχει υποχρεωτική περιφερειακή ε, προμήθεια. Αυτά θα πρέπει να, ε, οι τα θα πρέπει να από τις εθνικές αρχές, ε, οι οποίες έχουν το σωστό εξοπλισμό και θα πρέπει να αντιστοιχούν στις διαφορετικές γεωγραφικές συνθήκες κάθε κράτους, στις καταναλωτικές συνήθειες και στην διαμορφώση του δικτύου. Πρέπει να υπάρχει συνοχή με το στόχο δημιουργίας μιας πανευρωπαϊκής αγοράς και να υπάρχουν συνθήκε ε, ανταγωνισμού και αυτέ οι αλλαγέ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πρέπει μάλλον να συζητήσουμε πώς η τιμή θα αντικατοπτρίζει την ε, προσφορά και τη ζήτηση. Αν το αλλάξουμε αυτό θα πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας ε, το κοινό καλό. Αλλιώς τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Θα είναι δύσκολο να διασφαλίσουμε επενδύσεις, ειδικότερα αν θέλουμε να υποστηρίξουμε την καινοτομία και την καθαρή ενέργεια. Ε, θα είναι δύσκολο να έχουμε επενδύσεις ε, για παραγωγή και δημιουργία δυναμικότητας. Τώρα ο καταμερισμός κατά προτεραιότητα και οι καινοτομίες ε, είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την καινοτομία και τους σχετικούς πόρους, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να δημιουργήσει τεράστιες τρευλώσεις στην αγορά. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάποια εξισορρόπηση εδώ και συμφωνώ με την πρότασή σας επ' αυτού. Τώρα, Όσον αφορά τις εξαιρέσεις από την ευθύνη εξουσορρόφησης, αυτό μπορεί να αποτελέσει διακριτική μεταχείριση για όσους είναι υπεύθυνοι ε, από άψη εξουσορρόφησης, οπότε θα πρέπει να το σκεφτούν πολύ προσεκτικά. Όλοι οι φορείς της αγοράς θα πρέπει να υπόκειται στις ίδιες συνθήκες και να μην υπάρχει προτιμησιακή ε, μεταχείριση ε, ε, εκτός αν μπορούμε να καθορίσουμε, να εξηγήσουμε το αποτέλεσμα ενός τέτοιου μέτρου. Ε, οι προτάσεις μας πάντως ε, γενικά συμφωνούν μεταξύ τους. Στη συνάντηση που θα κάνουμε θα συζητήσουμε και περαιτέρω. Ευχαριστούμε κυρία Μπισνιεύσκα. Dziękuję bardzo Szanowni Państwo. Na wstępie chcę podziękować Panu. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο συνάδελφο για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Και έρχομαι τώρα στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμφωνούμε με τον στόχο και με μεγάλο αριθμό από τις προτάσεις που υποβάλλει η Επιτροπή. Δηλαδή, πράγματι χρειάζεται να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η αγορά ενέργειας και να ενταχθεί σε αυτό το ε, σύστημα ενέργειας ε, να ενταχθούν οι ανανεώσιμες πηγές. Δεν θα πρέπει να βλέπουμε τις ΑΠΕ σαν ένα βάρος, σαν μια δυσκολία. Αντιθέτως, είναι εξαιρετικά σημαντικές γιατί και μειώνουν το κόστος της ενέργειας και μας βοηθούν να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά βέβαια λαμβάνοντας υπόψη τις τροπικές ιδιαιτερότητες. Ε, για να γίνει λοιπόν αυτό με τρόπο αποτελεσματικό θα πρέπει να δώσουμε στα κράτη-μέλη τα εργαλεία που χρειάζονται. Πιο συγκεκριμένα να έχουν τη δυνατότητα να, να ε, επιλέγουν εκείνα, τα κράτη-μέλη δηλαδή, το ενεργειακό μείγμα που αντιστοιχεί στις ε, πηγές που έχουν στη διάθεσή τους και στις ιδιωτερότητες της κάθε χώρας πρέπει λοιπόν σε αυτόν τον τομέα να είμαστε προσεκτικοί. Δεν χρειάζεται να υπάρξει μία ε, μεταφορά αρμοδιοτήτων και να αρχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ε, τέτοιου τύπου αρμοδιότητες που δεν τις αντιστοιχούν, δεν τις αναλογούν. Ε, κατά την άποψή μου, αυτό είναι το πιο ευαίσθητο σημείο όσον αφορά τη ρύθμιση των στόχων για τις εκπομπές του του άνθρακα ανά κιλοβατόρα. Ε, έχουμε ήδη κανόνες για αυτά που, λειτουργούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια εβδομάδα πριν τη δημοσιοποίηση του προσχεδίου έλαβε μια απόφαση σε πολύ ψηλό επίπεδο εσωτερικά, χωρίς όμως να αξιολογήσει τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει αυτή η απόφασή της όσον αφορά τα όρια για το διοξίδιο του άνθρακα δεν θέλω να μπω στη συζήτηση του ότι επιδιώξεις μπορεί να κρύβονται από πίσω, αλλά πρέπει αυτούς τους μηχανισμούς και αυτά τα όρια να τους συμφωνούμε με τρόπο πραγματιστικό ε, που να προασπίζει το περιβάλλον χωρίς να επισέρχονται άλλα συμφέροντα σε αυτή τη συζήτηση. θέσαμε το ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν λάβαμε ικανοποιητική απάντηση ε, για το γιατί αυτό το όριο των 150 γραμμαρίων αλλά κιλοβατόρα εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα ε, προστατεύει το περιβάλλον πιο αποτελεσματικά από το όριο που είχαμε μέχρι τώρα. γνωρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει μια δέσμευση όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα των αερίων του θερμοκηπίου και μετά κάθε κράτος μέλος επιλέγει πώς θα συνεισφέρει στον στόχο αυτό. Ε, θα μπορούσε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο των κρατικών επιχορηγήσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πιο αποτελεσματικές ε, όμως δεν θα πρέπει να λάβουμε μέτρα τα οποία θα διακινδυνεύσουν την ενεργειακή ασφάλεια ορισμένων χωρών. Υπάρχουν χώρες όπως η δική μου, όπως η Πολωνία, που συνεχίζουν να, συνεχίζουν να εισάγουν φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Λέγεται ότι το TSO θα είναι ένα εργαλείο που θα βοηθήσει στην μείωση των εκπομπών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρξει ε, πρόβλημα στο κοινωνικό επίπεδο, να μην αυξηθεί υπερβολικά η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας ε, για τους καταναλωτές. Έχουμε ταυτόχρονα στόχους που έχουν θέσει οι εθνικές ε, κυβερνήσεις, όπως για παράδειγμα η κυβέρνηση της Πολωνίας, για τον εξηλεκτρισμό των μεταφορών. Ε, δεν αμφιβάλλω ότι ο εισηγητής είναι ένα λογικό άνθρωπο, αλλά ίσω να μην γνωρίζει σε βάθο την, κατάσταση σε ορισμένα κράτη-μέλη. Ένα άλλο στοιχείο που με ανησυχεί είναι ότι αυτά τα όρια τίθενται χωρί να προβλέπεται μεταβατική περίοδο. Σα δίνω κάποια στοιχεία λοιπόν τα οποία ελπίζω ότι θα βοηθήσουν να έχουμε πιο πιο, πιο επικοδομητική συνεργασία τις επόμενες εβδομάδες, έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση να μπορεί, που να ικανοποιεί όλα τα κράτη-μέλη. Κάθε κράτος μέλος να μπορεί να επιλέγει όπως το επιθυμεί εκείνο την ενεργειακή του πολιτική ε, για το μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Γιαταμάκη. Thanks. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Καρολίνα Πάντσα, της Κιώδης για την Άλντε, που δεν είναι παρούσα σήμερα, με παρακάλεσε να σας ε, υποβάλω τις εξής παρατηρήσεις. Σας διαβάζω λοιπόν το κείμενό της. Πρώτα απ' όλα, καλώς ορίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αποτελεί πολύ καλή βάση, διατυπώνει λογικές προτάσεις. Ευχαριστούμε τον συγκητή για την γνωμοδότησή του. Με πολλά σημεία μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ιδιαίτερος καλωσορίζουμε τις θέσεις του επί του εισηγητή ως προς τις, ε, τη διασυνδεσιμότητα για την, ε, και τη σημασία της για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Επίσης, συμφωνούμε με τις προτάσεις του εισηγητή για το μηχανισμό δυναμικού που πρέπει να στηρίζεται σε διαφανή κριτήρια και να μην αντιστρατεύεται του ενεργειακού και περιβαλλοντικού στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε κάποια μέτρα για την ενίσχυση των εξή διατάξεων. Πρώτα απ' όλα θέλουμε περαιτέρω να υποστηρίξουμε το ρόλο τη διασυνδεσιμότητα. Η υπερσυνοριακή συνδεσιμότητα αυτή τη στιγμή δεν εξυπηρετεί επαρκώς την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την αντιμετώπιση των ενεργειακών θυλάκων σε ορισμένε ε, περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι κάθε κράτος, κράτος μέλος θα πρέπει να φτάσει σε ένα επίπεδο διασυνδεσιμότητος που θα ισοδυναμεί με 10% τουλάχιστον με, την με το στιγμίο δυναμικό παραγωγής έως το 2020 για να προχωρήσουμε σε ένα πιο φιλόδοξο επίπεδο έω το 2030. Δεύτερον, Η αποθήκευση ενέργειας, πιστεύουμε, μπορεί να διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο για όλο το σύστημα, όχι μόνο περιορίζοντας ε, την, ε, τις μικροδιακοπές ε, στην παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αλλά εξασφαλίζοντας και τη δυνατότητα του πολίτη να <clears throat> μετατρέπεται σε παραγωγό ενέργειας και όχι μόνο σε καταναλωτή πράγμα το οποίο φαίνεται δύσκολο αυτή τη στιγμή. Η αποθήκευση μπορεί να διαδραματίσει πολύ πιο κεντρικό ρόλο στον κανονισμό δηλαδή. Τρίτον, για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση θεωρούμε ότι τα κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν ε, ακόμη επιτύχει τους ε, στόχους για ανανεώσιμες πηγές ε, θα πρέπει να προσυλλοθούν σε αυτό το στόχο και να τον τηρήσουν. Εν τέλει, θεωρούμε ότι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, οι μηχανισμοί θα πρέπει να, ε, δυναμικού θα πρέπει να στηρίζονται σε, ένα, σε μια αξιολόγηση συνεπειών με ε, υγιή βάση αξιολόγησης και με κριτήρια επιλεξιμότητας για τους παρόχους δυναμικού και βεβαίως περιμένουμε και προσβλέπουμε στην περαιτέρω συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος, κύριε Κίλλωναν. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή του δουλειά. Πάντα βέβαια παραμένει η δαμόκλος πάθη της κλιματικής αλλαγής. Για το κείμενο συγκεκριμένα. Για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία η θέση του πολίτη, του καταναλωτή. Η ενέργεια δηλαδή ως υπηρεσία είναι για μας κύριο σύνθημα. Γι' αυτό πρέπει να ακούσουμε τη γνώμη του καταναλωτή, του πελάτη. Για δικό του λογαριασμό πρέπει να λειτουργεί καλά η αγορά, να προχωρεί. Και σημειώνουμε ότι γίνονται πολλές επενδύσεις αυτή τη στιγμή στην ενέργεια σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, η ενεργειακή ένδυα παραμένει σημαντική πρόκληση. Δεν έχουν επαρκή πρόσβαση σε ενεργειακές πηγές όλοι οι πολίτες. Πρέπει να ε, επενδύσουμε σε ευέλικτες λύσεις. Πρέπει επίσης να μας απασχολήσουν δυνατότητες χρηματοδότησης που θα επιτρέπουν στον κάθε πολίτη να αξιοποιεί νέες λύσεις, καινοτόμες λύσεις, δυνατότητες που υπάρχουν ή που μπαίνουν στην αγορά. Χρειάζονται δηλαδή λύσεις ευφύης, χρειάζεται χτίσιμο πάνω στις λύσεις αυτές, καλές υπηρεσίες για τον καταναλωτή, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Τα νοικοκυριά, οι καταναλωτές πρέπει να είναι δηλαδή σε θέση να ωφελούνται από κάθε καινούριο προϊόν που μπαίνει στην αγορά, χωρίς αυτό να επιβαρύνει το λογαριασμό του ηλεκτρικού. Και πρέπει να δούμε τι μένει ακόμα να κάνουμε, τι πρέπει ακόμα να κάνουμε για τη βελτίωση της δεσιμότητας. Πρέπει να φτάσουμε δηλαδή σε ένα σημείο κατά το οποίο θα μπορούμε ισότιμα να μεταχειριζόμαστε κάθε τρόπο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ε, ταυτόχρονα να εξασφαλίζουμε την προμήθεια, τη σταθερότητα της προμήθειας σε ενέργεια. Ασφάλεια προμηθειών δηλαδή. Χρειαζόμαστε ασφαλώς περισσότερη εμπειρία για διαφορούς νέους τύπους ε, παραγωγής ε, ηλεκτρικής ενέργειας πριν φτάσουμε στην ε, ανέγερση μεγάλων ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων, γιατί βέβαια δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, να ξέρουμε επακριβώς τι κόστος, συνέπειες, αποδοτικότητα κτλ. μπορεί να προκύψει. Εμεί στις χώρες ε, του Βόρειου Αρκτικού Κύκλου έχουμε ένα σύστημα που φέρνει αποτελέσματα ικανοποιητικά με συνεργασία μεταξύ διαφόρων τομέων που ίσως μπορούν να αποτελέσουν και πηγή έμπνευσης για άλλες περιοχές της Ευρώπης. Thank you, Mr. Chair. Uh, first... Uh, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θέλω καταρχάς να καλωσορίσω την έκθεση του κύριου Μπέλετ. Συμφωνούμε σε πολλά σημαντικά θέματα. Κατά το σχεδιασμό όμω αυτού του νέου συστήματος για την επόμενη δεκαετία πρέπει να έχουμε μετρήσιμους στόχους. Πρώτα απ' όλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει Συμφωνία των Παρισίων. Εμείς έχουμε πει ότι θέλουμε να σταθούμε πρωτοπόροι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην αποδοτικότητα. Επίσης, δεύτερο και πολύ σημαντικό, οι πολίτες πρέπει να αποτελέσουν το επίκεντρο της ενεργειακής μετάβασης και έτσι το πακέτο θα πρέπει να εξασφαλίσει και ενέργεια σε καλές τιμές για τον καταναλωτή αλλά και καλές τιμές ενέργειας για την βιομηχανική παραγωγή. Έχουμε κάποιες εκθέσεις, και τροπολογίες για την έκθεση, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή συνεργασία, όχι μόνο περιφερειακά διαχειριστικά κέντρα ή λειτουργικά κέντρα, επιχειρησιακά κέντρα καλύτερα, ROCs, ε, αλλά επίσης και κάτι ακόμη που έχουμε, συνήθως, που έχουμε λησμονήσει ως συνήθως, τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες. και εδώ θέλω να σταθώ για να σας παρουσιάσω τις ε, θέσεις μας. Έχουμε λοιπόν μιλήσει για τα 350 γραμμάρια ένα κιλοβατόρα όριο στις εκπομπές. Ωστόσο εδώ έχουμε και τα όρια που μας επιβάλλει η τεχνολογία, η τεχνολογική πρόοδος. Εάν μας λένε οι χειριστές, οι ε, οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγικές με τις τουρμπίνες ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για, και οι επενδύσεις περισσότερες για την ανάπτυξη καλύτερης ε, τεχνολογίας. Θα πρέπει αυτό να το κάνουμε και πρέπει να εξασφαλίσουμε στο δυνατόν καλύτερη ευελιξία στο σύστημα. Γιατί δεν αρκεί να έχουμε το δυναμικό ε, ως αποθεματικό, αλλά το δυναμικό σε δυνατότητα παραγωγής. Και οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουμε πιο φιλόδοξα επίπεδα και να αποστείλουμε ε, και μήνυμα προς τη βιομηχανία ότι κάποια στιγμή η αποθήκευση θα τερματιστεί. Γιατί έχει πάρει πλέον, ε, όχι εμπορικά, εμπορικές διαστάσεις, αλλά διαστάσεις επιστημονικής φαντασίας αυτή η ιστορία. Περιφερειακή συνεργασία. Υποστηρίζουμε την προσέγγιση της ισότιμης αντιμετώπισης των πόρων. Είναι σημαντικό σε εθνικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο να εξασφαλιστεί η συμφωνία στην κατεύθυνση αυτή. Και βεβαίως Θέλουμε να ανταποκριθούμε στις ε, προσδοκίες των πολιτών μας. Στο κέντρο της, ε, μεταβατη... της ενεργειακής μετάβασης πρέπει να ε, χθεί ο πολίτης και να ανοίξει χώρος για νέους φορείς με τον καταναλωτή στο δικαίωμα στην αυτοκατανάλωση, ιδιοπαραγωγή και προαγωγή της μετάβασης που δεν υπάρχει, εκεί όπου δεν υπάρχει. και που μπορεί στα επόμενα χρόνια να εμφανιστεί. Προτεραιότητα εξυπηρέτησης. Θέλουμε να είμαστε λοιπόν ηγετική δύναμη στις ανανεώσιμες πηγές, να επιτύχουμε τους στόχους των Παρισίων και ως εκ τούτου πρέπει να μας απασχολήσει το σύστημα διανομής και εξυπηρέτησης χρειάζεται μια αξιολόγηση της κατάστασης. όχι αναδρομικό, με προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση για τα νέα προϊόντα, αλλά όχι αναδρομικά. Και αξιολόγηση συνεπειών. όταν συμμετέχουν στην αγορά. Και βεβαίω προσβλέπουμε σε πολύ καλή συνεργασία με τον εισηγητή στην ολοκλήρωση των γράφων. Thank you. Um, next speaker, Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να υποστηρίξω τον υποπλετών ε, εισηγητή είναι σαφές ότι η αγορά ηλεκτρική ενέργειας πρέπει να είναι πιο ευέλικτη γιατί πρέπει να ενσωματώσουμε τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και να υπάρχει πιο δυναμική κατανάλωση από του πολίτε μα. Ε, είναι πολύ καλή λοιπόν η ισορροπία που έχει επιτύχει ο εισηγητή μα. Θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να υλοποιήσουν μηχανισμού δυναμικότητα, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ασφάλεια του εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια αλλά Εκτιμώ ότι αυτοί οι μηχανισμοί δεν πρέπει να υπόκειται σε μία μελέτη επάρκειας. Χρειαζόμαστε ένα μακροχρόνιο όραμα. Οτιδήποτε εμποδίζει αυτό το μακροχρόνιο όραμα πιστεύω θα αποτελέσει εμπόδιο. Όσον αφορά τι ανανεώσιμε πηγές ενέργειας, εξελίσσονται όλο και περισσότερο, αυτό είναι καλό. Αλλά θα ήθελα ε, προτεραιότητα εισαγωγή στο δίκτυο να ε, να προτεραιότητα να δοθεί στις μικρές εγκαταστάσεις οι οποίες χρειάζονται ακόμα υποστήριξη, ε, μικρές θαλάσσιες εγκαταστάσεις. Ε, πρέπει να συνεχίσουμε να τους παρέχουμε αυτή την προτεραιότητα. Όσον αφορά τη δημιουργία περιφερειακών ε, λειτουργικών κέντρων, καλή ιδέα, αλλά και εκεί δεν πρέπει τα κέντρα αυτά να καταργούν τη δυνατότητα για τους TSO να ελέγχουν την ισορροπία ε, της, του εφοδιασμού. Οπότε πιστεύω ότι η μεταφορά της ανάλυσης ε, των αναλυτικών κέντρων σε αυτά τα περιφερειακά κέντρα είναι καλό πράγμα, αλλά πρέπει οπωσδήποτε οι λειτουργικές ε, εργασίες να μην μεταφερθούν και αυτές, γιατί εκεί θα έχουμε πρόβλημα, θα βρίσκεται αλλού θα λαμβάνεται αλλού η απόφαση και αλλού θα υπάρχει ευθύνη. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε λοιπόν. Αυτά είναι τα λίγα στοιχεία με τα οποία θα ήθελα να συνεισφέρω και εγώ στη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γκροστέτ. Ο κύριος Λίζα. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ τον Ρεβομπέλετ για την πρόταση. Θέλω και, εκ μέρους του και τον κύριο Χάριν να ευχαριστήσω που είναι ο αρμόδιος εκ μέρους της Ήτρε για τη σύνταξη της μομοδότησης. Χρειαζόμαστε λοιπόν στην ενέργεια και γνήσιο ανταγωνισμό και καινοτομία. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι εργάζονται ακαταπώνητα για να βρουν νέε λύσεις ε, για την εξίσωση της ε, ενεργειακής αποδοτικότητας, διαφόρων ε, πηγών. Έχω, παραδείγματι, επικοινωνήσει με ένα μεγάλο παραγωγικό αλουμινίου της Γερμανίας, που είναι καταναλωτής του 1% της ε, γερμανικής, ε, στη Γερμανία παραγόμενης ενέργειας, ο οποίος είναι σε θέση, είναι υποχρεωμένο να σταματήσει την ε, παραγωγή του τη στιγμή που βλέπει κάποια ανομαλία στην παραγωγή ενέργειας για να μην, ε, στην διάθεση μάλλον της ενέργειας για να μην ε, κινδυνέψει το σύστημα παραγωγής. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι μπορούμε να τα αφήσουμε όλα στην αγορά. Χρειάζεται ένα στρατηγικό αποθεματικό με όσο δυνατόν λιγότερη παρέμβαση από δική μας πλευράς, δηλαδή η αγορά μεν πρέπει να λειτουργήσει ελεύθερα. Αυτό που δεν κατάλαβα από την κυρία Βυσνιέσκα, γιατί άκουσα να λέει ότι είναι αρμοδιότητα η ιστορική αγορά των κρατών μελών. Ε, πρόκειται για οξύμορο ασφαλώ, διότι η ιστορική αγορά είναι πυλώνας Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, μπορεί να ρυθμίζουν την ιστορική του αγορά ενέργειας στα κράτη-μέλη, αλλά όχι την ιστορική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωση. Και αν πάμε προς τα εκεί θα γίνουν όλα πιο ακριβά. Η πρόταση για τα 150 γραμμάρια της Επιτροπής είναι θετική για μένα. Δεν την έχει αμφισβητήσει ο κύριος Κάρενς. Αλλά φαντάζομαι ότι σημαίνει πως πρόκειται για ένα στρατηγικό απόθεμα και όχι για αγορά δυναμικού. Επίσης καλωσορίζω την πρόταση του Ιβο Μπέλετ για την ε, εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα. Νομίζω ότι ε, αυτό δεν πρέπει να προχωρήσει έτσι, γιατί θα πρέπει να αποδείξουν την αξία τους οι ανανεώσιμες πηγές μέσα από την αγορά. Ίσως να φανεί ότι χρειαζόμαστε για ένα διάστημα ακόμα την ε, ε κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση. Ο κύριος Πάλτσο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Η ρύθμιση της τουρκικής αγοράς είναι βέβαια καυτό θέμα. Είναι πολύ σημαντικό να ορίσουμε ποιοι είναι οι τομείς, οι στόχοι και οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποιες αρμοδιότητες παραμένουν στα χέρια των κρατών μελών. Είναι νομίζω χαρακτηριστικό το ότι 8 ε, εθνικά κοινοβούλια διατυπώνουν γνωμοδότηση σε αυτή την έκδοχη. Κοινοβούλια τα οποία φρονούν ότι παραβιάζεται από τις νέες αυτές προτάσεις η αρχή της επικουρικότητας. Το Ουγγρικό Κοινοβούλιο, παραδείγματι με τη γνωμοδότησή του, δηλώνει ότι Ο προσδιορισμός του δυναμικού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας και ε, το άρθρο 23 παραβιάζει, περιστέλει τη δυνατότητα των κρατών μελών να προσδιορίσουν από μόνο τους το ενεργειακό μείγμα. Επίσης, τομείς διάφοροι και συγκεκριμένοι, όπως και αρμοδιότητες διάφορες και συγκεκριμένες, παρουσιάζοντας ε, αρμοδιότητες και τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ πρόκειται για δραστηριότητες νομοθετικές των κρατών μελών. Επίση, η γνωμοδότηση του Γκρικού Κοινοβουλίου μα λέει ότι έχουν τα κράτη-μέλη στα ε, διάθεσή του μέτρα, μέσα μάλλον εργαλεία προστασία των καταναλωτών. Και περιορισμού της ε, ενεργειακής ένδυας. Ο προσδιορισμός των τιμών σε επίπεδο αγοράς, σε ποιο βαθμό όμως περιορίζει δηλαδή το μελών για προσδιορισμό αυτών των τιμών. Σας ευχαριστώ. Ακούσαμε όλους τους ε, σκιώδης και τον εισηγητή. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν προφέρω το σωστά το όνομά σας, κύριος Βαχανχάμστερν. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία να εκφράσω τις πρώτες αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτή τη συζήτηση τη σημερινή. Καλωσορίζουμε ορίζουμε όλες τις απόψεις που εκφράστηκαν, όλες αυτές τις συνεισφορές των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να σας εξηγήσω ορισμένε από τις πρώτες μας αντιδράσεις όταν διαβάσαμε τις προτινόμενε τροπολογίες. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να υπενθυμίσω ότι ο λόγος για τον οποίο υποβάλλει αυτήν την πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δύο στόχοι ουσιαστικά. Πρώτα απ' όλα να εξασφαλίσουμε ότι η αγορά θα είναι έτοιμη να υποστηρίξει τις ΑΠΕ με άλλα λόγια να δώσουμε κίνητρα για αυτή την ευελιξία και να εξασφαλίσουμε ότι όλα, όλα, όλα και επιχειρήσεις οι μπορούν να, αξιοποιήσουν αυτή την ευελιξία θα είναι έτοιμες να μπουν στην αγορά και μετά να ε, εξασφαλίσουμε ότι η ενεργειακή μετάβαση θα γίνει με τρόπο οικονομικά αποτελεσματικό. Πριν δέκα χρόνια συζητούσαμε για τις ΑΠΕ σαν να ήταν μια, γινόταν μια συζήτηση καταγγελτική, σαν ήταν άσπρο μαύρο. Σήμερα βλέπουμε ότι εισάγονται στην αγορά σταδιακά και μέχρι το 2030 προβλέπεται ότι το 60% της ενέργειάς μας θα προέρχεται από ΑΠΕ. Βέβαια. Αυτή τη στιγμή έχουμε εξαιρέσεις για τις ΑΠΕ στο ρυθμιστικό πλαίσιο, οι οποίες δεν έχουν πλέον ε, νόημα. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επανεξετάσει την πρόταση της Επιτροπής, η οποία έχει μια συγκεκριμένη ισορροπία. Προσπαθούμε τα κράτη-μέλη να ε, υποστηρίξουν τις ΑΠΕ και μόνο εκεί που χρειάζεται να υπάρχουν εξαιρέσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο για το ενδιακό του μείγμα δηλαδή. Η πρόταση της Επιτροπής εξάλληψε ουσιαστικά από το τρίτο πακέτο για τα ενεργειακά πυρήνα. Τη δυνατότητα μεταφοράς επιχορηγήσεων, εάν ακούσαμε σωστά τον ομιλητή, χωρίς αυτό να δημιουργήσει προβλήματα στην διασύνδεση. Το ζήτημα λοιπόν που τίθεται είναι πώς μπορούμε να διευκολύνουμε και πάλι αυτές τις πρωτοβουλίες και με ποιες προϋποθέσεις. Ποιες λοιπόν θα πρέπει να είναι οι νέες προϋποθέσεις που θα εισαγάγουμε για τη χρήση του εισοδήματος συμφόρησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν καλοβλέπει τα εθελοντικού χαρακτήρα κριτήρια, τα οποία θα είναι πολύ δύσκολο να προσαρμοστούν στις εθνικές ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους. Θα ήταν χρήσιμο να μην ξεχνάμε ότι η διασύνδεση δημιουργείται απλώς με τους ε, αγωγούς, αλλά το ζήτημα είναι να υπάρχει και διαθέσιμη ενέργεια στο άλλο άκρο της ε, διασύνδεσης, έτσι ώστε να μπορεί να μεταφερθεί. Η μεταφορά ε, ηλεκτρικής ενέργειας επίσης έχει ένα κόστος. Η πρότασή μας λοιπόν είναι πρώτα απ' όλα κατά προτεραιότητα η το, το εισόδημα συμφόρηση να χρησιμοποιείται για να βελτιωθούν οι διασυνδέσεις και δεύτερον, να συμπεριληφθούν στα κριτήρια και ορισμένα κόστη που σήμερα δεν συμπεριλαμβάνονται. Κάτι το οποίο θα βελτιώσει τη διασύνδεση μέχρι και το επίπεδο του, του να είναι διαθέσιμη για την χρήση από τον καταναλωτή αυτή η, ενέργεια που προέρχεται από της, τη διασύνδεση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως σας είπα, τονίζει τη σημασία των ΑΠΕ. Επίσης θεωρεί ότι η αγορά έχει τις δυνατότητες να χρηματοδοτήσει αυτή την κοινοτομία πιο αποτελεσματικά. Σήμερα σε διάφορα είδη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχουν επιδοτήσεις οι οποίες οδηγούν σε, μια, σε υπερβολικό δυναμικό, σε υπερβολική παραγωγή. Πρέπει λοιπόν να εισάγουμε στο σύστημα μας το εξή. Ότι για τις επιδοτήσεις θα λαμβάνεται υπόψη το δυναμικό μόνον όταν αυτό είναι απαραίτητο. Και επίσης ότι θα υπάρχει ένα όργανο σε κάθε κράτος μέλος που θα κάνει αυτή την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση αυτή πρέπει βέβαια να λαμβάνει υπόψη της, τις σε εθνικό επίπεδο, ναι. Αλλά κάτι που ίσως δεν ήταν πολύ ξεκάθαρο για μένα όταν διάβασα τις προτάσεις τροπολογιών είναι ότι είχε τεράστια σημασία να χρησιμοποιείται μία ενιαία αναρμονισμένη μεθοδολογία από ένα, από ένα ε, κεντρικό όργανο για να γίνονται αυτές οι εξελογήσεις, το οποίο με φέρνει και στο όριο των 150 γραμμαρίων ένα κιλοβατόρα. Ε, γνωρίζω ότι το ζήτημα αυτό προκαλεί διχογνωμία, δεν είναι εύκολο. Όμως δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε όσον αφορά ε, τα αποτελέσματα, τις επιπτώσεις που θα έχει το μέτρο αυτό. Έχουν διεξαχθεί μελέτες από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που θα σας παράσχουμε ένα αυτό το χρόνο για να διευκολύνσουμε τη συζήτηση και οι οποίες έχουν μελετήσει την οικονομική αποδοτικότητα αυτού του συγκεκριμένου μέτρου και γενικότερα μέτρων τα οποία θέτουν συγκεκριμένα όρια ανάλογα με τη δυναμικότητα του, του, του, του, του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ε, μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση, δεν θα πω σε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ. Όσον αφορά τα περιφερειακά κέντρα, τα ΡΟΚ, η πρόταση της Επιτροπής δεν είναι κάτι το τελείως καινούριο, είναι μια εξέλιξη ε, αυτού που ήδη συμβαίνει, της περιφερειακής συνεργασίας που ήδη υφίσταται. Νομοθετείται αυτό, ωστόσο παραμένει στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών και των TSO να βρουν τα, το συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας αυτών των περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων. και να διευκρινίσουν τροποντινά ποιο συνεργάζεται με ποιον. Δεν προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από πάνω προ τα κάτω να επιβάλλει κανόνε σε αυτόν τον τομέα. Αντιθέτω. Σε δεύτερο γενή νομοθεσία, κάτι το οποίο έχουμε τη δυνατότητα πια να υιοθετήσουμε με το τρίτο πακέτο για την ενέργεια, θα ε, διευκρινιστούν και οι τεχνικές λεπτομέρειες θα σας ζητούσα να θεωρήσετε τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα τα ΡΟΚ ως ένα θεσμικό όργανο το οποίο θα εξασφαλίζει την υλοποίηση και την τήρηση των κανόνων που συμφωνούμε. Γι' αυτό έχει αλλάξει και η διατύπωση πλέον δεν, ε, και η νομική μορφή. Δεν είναι, πρόκειται πλέον για απόφαση της Επιτροπής αλλά για σύσταση. Αυτό έχει τη σημασία του. Γιατί υιοθετώντα την νομική ε, μορφή τη ε, σύσταση κάνουμε ένα βήμα προ τα πίσω σε σχέση με το σημερινό νομικό καθεστώς. Είναι ε, ένα θέμα σημαντικό και πρέπει να δούμε αν πραγματικά αυτό επιθυμούμε. Στη συζήτηση για τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα μερικές φορές ακούγεται η άποψη ότι είναι κάτι του καινούριο. Δεν ισχύει αυτό. Πρόκειται για μια αποκριστάλλωση μια συνεργασίας που ήδη προβλέπεται στη σημερινή νομοθεσία και πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο και για τη λειτουργία τους. Τώρα θα δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου ε, που θα διευκρινίσει ε, επιπλέον στοιχεία της Ευχαριστώ. Ονομάζομαι ρωσάντε και έχω δύο βασικά θέματα. Το ένα αφορά τις προτάσεις για τη δημιουργία, για τη διαμόρφωση των τιμών. Είναι σαφές ότι στην πρότασή μας θέλουμε οι τιμές να διαμορφώνονται βάσει της ε, ζήτησης και της προσφοράς. Αυτό δεν είναι γενικό ζήτημα. Μπορεί να υπάρξουν και εξαιρέσει. Μπορεί να υπάρχουν σε εξαιρετικές περιπτώσεις τιμές ε, ε, βάσει ε, προσφορά και ζήτηση και βάσει τη αγορά ώστε να υποστηρίζουν την καινοτομία. Τώρα για τους TSO ε, υπάρχει μια πρόταση να συμπεριλαμβάνεται όλη η ΔΕΣΟ και να υπάρξει σωστή μεταξύ των μελών ε, ε της νέας οντότητας αυτής ε, και του κράτους μέλους. Αλλά εμείς θεωρούμε ότι η Ένωση του Φυσικού Αερίου δεν πρέπει να συμμετέχει ότι θεωρούμε ότι δεν θα λειτουργήσει όλο αυτό. Θα στείλουμε εμεί σχόλια γι' αυτό, ώστε να μην υπάρξουν μεγαλύτερε δυσκολίε για να λειτουργήσει αυτή η οντότητα των TSO. οι TSO υποστηρίζουν το 90% περίπου των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια σε ορισμένα κράτη-μέλη. Οπότε υποστηρίζουμε τη συνεργασία μεταξύ TSO. Αυτή η νέα οντότητα, λοιπόν, αυτό ο νέο οργανισμό δημιουργήθηκε ακριβώ για αυτό. Για να ενισχύσει τη συνεργασία με τους, ε, μεταξύ των TSO. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε στον κύριο Μπέλετ, στον εισηγητή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, θα είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομος. Ευχαριστώ όλους τους κοιόδης και όλους τους συναδέλφους. Πολλές πληροφορίες ακούσαμε, πολλές απαντήσεις θέλω να δώσω, θα προσπαθήσω να τις συνοψίσω. Κύριε Πότσα, φυσικά ναι, έχουμε συμφωνήσει ήδη από σήμερα το πρωί να κάνουμε μια όμορφη συνάντηση με καφεδάκι την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσουμε περαιτέρω τα όλα θέματα και να προσπαθήσουμε να κάνουμε να συγκλίνουν οι δύο εκθέσεις. Ε, για τις απαντήσεις σας για το νέο ζώο που έτσι όπως το ονομάσαν ε, οι Κομισιόν, ε, οι περιφερειακές οργανώσεις αυτές, ναι πρέπει να το εξετάσουμε πιο προσεκτικά. Δεν θέλουμε φυσικά να υπονομεύσουμε το υπάρχον και εκτιμένο, αντιθέτως θα έρθουμε σε επαφή και θα βρούμε μια πολύ καλή λύση. Ο καταμερισμός κατά προτεραιότητα, Παύελ, ε, ναι, από όσο κατάλαβα, δεν είστε απόλυτα ευχαριστημένος με αυτό, αλλά θα πρέπει να το δούμε παρα παρακάτω. Μιλήστε για ισορροπία, θα βρούμε μια λύση γι' αυτό. Κυρία Βυσνιεύσκα, είστε εδώ, ναι. Μπορώ, πιστεύω να σας πείσω, κυρία Βυσνιεύσκα, ότι όχι μόνο έχουμε επαφή με ε, την κατάσταση στη δική μου χώρα αλλά ήρθα σε επαφή και με πολλούς συναδέλφους ε, πριν από την κατάρτιση αυτής της ε, γνωμοδότησης οπότε γνωρίζουμε απόλυτα και βάσει των πληροφοριών του Αντρέ και άλλων ε, συναδέλφων από την Πολωνία και από άλλε χώρε τη Ανατολική Ευρώπη για το πόσο ευαίσθητο είναι το θέμα αυτό σε ορισμένα κράτη-μέλη. Και επιτελεί. Ε, ε, αντιδράσατε. Ναι, φυσικά δεν θέλουμε να παρέμβουμε στο ενεργειακό μείγμα. Σίγουρα από τη εθνική αρμοδιότητα. Δεν είναι κάτι το οποίο εμεί θέλουμε να αφισβητήσουμε. Αλλά εδώ μιλάμε για την εσωτερική αγορά και για τι αλληλεπιδράσει εντό της ε, εσωτερικής αγοράς χωρίς να παρεμβαίνουμε στο ενεργειακό μείγμα. Θέλουμε να έχουμε μια κατάσταση όπου όλοι θα κερδίζουν συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών. Οπότε η ασφάλεια εφοδιασμού είναι ένα από τα βασικά μας θέματα. Ε, η ασφάλεια εφοδιασμού και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν μπορούμε να τα διαχωρίσουμε. Ε, αλλά ακούμε τις ανησυχίες σας και φυσικά θα τις λάβουμε υπόψη η κυρία Γέτεν Μάκη. Αναφερθήκατε στην πτυχή της διασυνδεσιμότητας. Ο καθαμερισμός κατά προτεραιότητα, το priority dispatch που ανέφερε η κυρία Γκροστέτ ε, και ο κύριος Λίσερ, πολλοί συναδελφοί λένε ότι πρέπει να είναι προσωρινό. Δεν είναι πρόθεσή μα σε καμία περίπτωση να τον καταργήσουμε μέσα στα επόμενα χρόνια. Όπως ανέφερε και η Φρανσουάζ θα ληφθεί υπόψη Τώρα να μιλήσουμε για τα καινετόμα μικρά έργα που ε, εμφανίζονται στην αγορά. Εκεί ο καταμερισμός κατά προτεραιότητα ε, εξακολουθεί να αποτελεί μια καλή ιδέα. Οπότε δεν μπορούμε να τον αποκλείσουμε. Κύριε Κιλώνεν, ε, εστιαστήκατε στον καταναλωτή για το πώς θα τους βοηθήσουμε να δρουν έξυπνα. Φυσικά αυτός είναι από τους κύριους στόχους. Συμφωνούμε απόλυτα να ενθαρρύνουμε τους καταναλωτές να ε, ε, είναι αποτελεσματικοί ως προς το κόστος, είναι από τους κύριους μας στόχους αυτός. Ο κύριος αναφέρθηκε στο ότι ο μηχανισμός δυναμικότητας έχει να κάνει με ευελιξία και ότι πράγματι ορισμένα ε, εργοστάσια φυσικού αερίου θα μπορούσαν να ανανεωθούν σήμερα μέσω κάποιες καινοτόμια. Συμφωνώ με αυτή την πρόταση. Είναι μια από τις λύσεις που προτείνονται όσον αφορά το μηχανισμό δυναμικότητας. Ξέρεις τον κύριο Μπάλτσα, ε, αλλά νομίζω έχει φύγει. Μίλησε για την επικουρικότητα. Φυσικά όλοι συμφωνούμε ε, όσον αφορά την επικουρικότητα, αλλά επαναλαμβάνω, δεν ήταν πρόθεσή μας ε, να στραφούμε κατά των κρατών μελών ε, όσον αφορά την αρμοδιότητά τους σε θέματα ενεργειακού μείγματος. Ε, το θέμα εδώ είναι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, πώ θα τι παντρέψουμε με την, ενέργεια, με την ασφάλεια εφοδιασμού και αυτό που μα ανησυχεί κυρίω έχει να κάνει με τα αποτελέσματα αυτή τη αναδιοτύπωση στον καταναλωτή, στι εκπομπέ και στην ασφάλεια εφοδιασμού. Αυτό είναι που ανησυχεί τον κύριο Μπάλτσε και αυτό ανησυχεί και εμένα και αποτελεί κύρια μα προτεραιότητα. Αυτά είναι τα κύρια σημεία Υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ ε, απόψει, οπότε θα ανταλλάξουμε απόψει με του κοιόδη μέσα στι επόμενε ημέρε και εβδομάδε και αναμένουμε τα σχολεία σα. Ευχαριστώ. Ε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για αυτή τη συζήτηση, η οποία θα συνεχιστεί, είναι βέβαιο. Ε, προθεσμία για τις τροπολογίες η 10η Οκτωβρίου 11 το πρωί. Και θα ψηφίσουμε στην ΕΜΒΗ τον Νοέμβριο. 21 Νοεμβρίου. Ωραία. Πάμε στο τελευταίο σημείο της ημερησίας διαταξής σήμερα και αυτό έχει να κάνει με τις μέλισσες. Προοπτικές και προκλήσεις για τον τομέα μελισσοκομείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε το σχέδιο έκθεσης της κυρίας Ντορνανό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης που μου ανατέθηκε είναι πολύ σημαντικό για μένα. Η επιβίωση των μελισσών αποτελεί επίκαιρο θέμα, φλέγον επίκαιρο θέμα και αυτή είναι η μόνη γνωμοδότηση που θα δοθεί στην Επιτροπή Αγκρή, η οποία είναι επί της ουσίας αρμόδια. Την περασμένη εβδομάδα Μετέμεινε στην εκλογική μου ε, περιφέρεια στο γαλλικό παρατηρητήριο Μελισσών σε ένα βιότοπο ε, ειδικά αφιερωμένο για την έρευνα και την παρατήρηση και εγώ συζήτησα με μελισσοκόμους και ερευνητές στόχος των οποίων ήταν να επιλέξουν τις ε, πιο ανθεκτικές και παραγωγικές μέλισσες, να τις αναπαραγάγουν και να εκπαιδεύσουν τους γεωργούς να κάνουν το ίδιο. Αυτή η ανταλλαγή απόψε ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και με καθυσίχασε η όλη κατάσταση. Ο, θεωρώ ότι οι αποφάσεις του Κοινοβουλίου θα, έχουν, ε, θα σημαντικά και θετικά το μέλλον. Η γνωμοδότηση που παρουσιάζω σήμερα φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στη βασικά ερωτήματα που αφορούν το μέλλον του τομέα της μελοσοκομείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ ρώτησα από όλους επιστήμονες, ερευνητές και ειδικού για το θέμα αυτό Όσον αφορά τώρα το σχέδιο γνωμοδότησής μου, ε, το σχέδιο εκθεσή μου, ήθελα να επιμείνω ότι οι μέλισσε αποτελούν απαραίτητο στοιχείο της βιοπικιλότητας, ότι αποτελούν ε, αναντικατάστατη παγκόσμια κληρονομιά, διότι από αυτές εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η ζωγαμία, δηλαδή η επικονίαση μέσω των ζώων όσον αφορά την προβληματική της επιλογής των μελισσών επιτρέπει την αντοχή σε ορισμένε ασθένειε, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε να μελετάμε το σύνολο των κινδύων που σχετίζονται με την πτώχυνση του γενετικού, ε, της γενετικής ε, κληρονομιάς των ε, μελισσών, ειδικότερα των τοπικών ειδών. Πρέπει να δούμε και τα αποτελέσματα της γενικής χρήσης ζυζανιοκτώνων, ειδικότερα για τα μελιφόρα φυτά. Δεκάδες ε, πολίτες μας έχουν στείλει αναφορές ε, κάνοντας έκκληση μα γενική απαγορεύση των νεονικοτινοειδών. Πρέπει οπωσδήποτε να εισακούσουμε να εισακουστούν αυτές οι ανησυχίες και να εξετάσουμε τα αποτελέσματα. Διαπιστώσεις με διαφάνεια και πρόταση ε, οδών επίλυσης είναι αυτό που πρέπει να γίνει επιπλέον. Γι' αυτό υπογραμμίζω το ότι η ελεγχόμενη επικονίαση μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση της αρμονίας μεταξύ μελισσοκόμων και γεωργών και να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργιών τους. Εάν η επιβίωση του μελισσοκομικού τομέα πρέπει να αντιμετωπιστεί και όχι μόνο στο μέτωπο της παραγωγής αλλά και στο μέτωπο της ε, ε, εμπορικής διάθεσης. Απαιτούνται σημαντικά μέσα για να καταπολεμηθούν οι περιπτώσεις απάτης και του ανταγωνισμού, ε, ειδικότερα στις περιπτώσεις του νοθευμένου μελιού. Η επιβίωση των Ευρωπαίων μελισσοκόμων θα πρέπει να οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσαρμόσει τους στόχους ε, της κοινή γεωργικής πολιτικής ε, όπως τον πολύ αφισβητήσιμο στόχο της αύξησης της παραγωγικότητας. Πράγματι, η διαρκώς αυξανόμενη παραγωγή των καλλιεργειών ε, θα δημιουργήσει πρόβλημα ε, στην επιβίωση των μελισσών. Μετά από την επίσκεψη που έκανα στο Γαλλικό Παρατηρητήριο Μελισσοκομείας ήθελα να επιμείνω στο ρόλο της έρευνας για τις αιτίε ε, της μείωσης του προσδόκιμου ζωής των βασιλισσών. Κάτι που αποτελεί ανησυχητικό φαινόμενο. Θεωρώ σκόπιμο να υποστηρίξουμε με όλα τα δυνατά μέσα την ανάπτυξη βιολογικών φυτοφαρμάκων που δεν βλάπτουν τις μέλισσες ώστε να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατα των νέων οικοτινοειδών και της ε, που έχουν επαληθευμένη τοξικότητα για τις μέλισσες. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την εκπαίδευση και κατάρτιση των μελισσοκόμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της χρήσης δικτών επιβίωσης ε, των απικιών ε, βάσει μοντέλων που υπάρχουν ήδη. Τέλος, στο σχέδιο γνωμοδοτησή μου ζητούμε ενίσχυση των μέσων που διατίθενται για την καταπολέμηση της εμπορικής απάτης, η οποία επηρεάζεται με λισοκόμικά προϊόντα, ώστε να αντιμετωπίσουμε πραγματικά αυτά τα προβλήματα. Το να καταγγέλουμε προβλήματα χωρίς να παρέχουμε τα μέσα καταπολέμησής τους δεν έχει νόημα. Είμαι έτοιμη να απαντήσω σε ερωτήσεις και να ακούσω τι παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ εκ των προτέρων όλους όσους θα συμμετάσχουν. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, can... Ευχαριστώ πολύ. Σκιώδης τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για την παρουσίαση του θέματος. Δεν έχουμε χρόνο θα μιλήσω λοιπόν συγκεκριμένα για διάφορες προτάσεις, παράγραφοι 9 και 10, δομή και μετά περιεχόμενο, παράγραφος πρώτη. Στη διατύπωση βλέπω κάποιο πρόβλημα, ας το δούμε, μήπως θα έχει μετάφραση. Παράγραφος 2. Επιλογή επιζώτιων που πλήττουν την ε, μέλισσα. Και έτσι θα έλεγα όχι μάστιγες για την υγεία, να μην είμαστε και τόσο συναισθηματικοί, να μιλήσουμε πιο ουσιαστικά και αντικειμενικά. Παράγραφος 3. Λαμβάνει υπόψη ε, ε, μέτρα που έχουν ήδη αναλυφθεί για φυτοπροστασία και παρά είναι αυστηρή στη διατύπωσή τη. Η παράγραφος παριθμών 6 με προβληματίζει σε σχέση με τη διατύπωση και τους προσανατολισμούς. Δεν λαμβάνει υπόψη μη οικολογικής εστίασης, πρασίνισμα στην γεωργία και το καθεξής. Παράγραφος 8 φυτοπροστασία, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, που μπορούν να μας επιτρέψουν να βρούμε λύσεις στα προβλήματα. Για προϊόντα που έχουν αποδειχθεί επικίνδυνα και απαγορευθεί. Κατάρτιση για το μελισσοκόμμα βεβαίως, απολύτως απαραίτητη. Ε, πολλές φορές ε, ξεκινάει σαν χόμπι, σαν παρέργο, χωρίς γνώση και μπορεί να φέρει και προβλήματα αν δεν υπάρχει κατάλληλη κατάρτιση. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ όλη αυτή η ιστορία γιατί είμαι μεταξύ αυτών των βουλευτών που ασχολούνται πολύ με τα θέματα της ε, μελισσοκομείας ε, και η ε, ήμερη αλλά και η άγρια μέλισσα έχουν τεράστια σημασία για την επικονίαση. Ευχαριστώ. Πιαγκά. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ την εισηγήτρια. Ευτυχώ δεν είναι υπερβολικά μακροσκελή η γνωμοδότηση. Θέμα που συχνά μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα. Ωστόσο έχουμε έχουν επισημανθεί τα κύρια προβλήματα σε σχέση με τη διάρκεια ζωής των βασιλισσών και τα βιολογικά βιοκτώνα. Ο θέμητος ανταγωνισμός βεβαίως πρέπει να καταπολεμηθεί με το αλλοιωμένο μέλι. Το μέλι είναι ένα σαφώς προσδορισμένο φυσικό προϊόν με συγκεκριμένα συστατικά που ορίζονται από κανονισμούς με το τελευταίο του 2016 και είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί η ε, εμπιστοσύνη του καταναλωτή στο μέλι ως προϊόν. Πρέπει να είναι ο καταναλωτή ότι όταν παίρνει μέλι εισαγωγή από τρίτε χώρες θα είναι και αυτό καλή ποιότητα. Πρέπει λοιπόν να αποφεύγονται οι απομιμήσει και οι παραποιήσει με στόχο πάντα την προστασία του καταναλωτή. Σε ένα σημείο όμω θα ε, πω ότι διαφωνώ διότι δεν πιστεύω ότι ο θάνατος των μελισσών ε, προξενείται μόνο από τα χημικά ζυζανιοκτώμα, γιατί και ζυζανιοκτώνα, γιατί και στην βιολογική καλλιέργεια συμβιώνονται θάνατοι μελισσών. Με ακόμα ευνοϊκότερη υποτίθεται ε, σύσταση του περιβάλλοντος για την Μέλισσα, βλέπουμε πάλι σημαντικούς αριθμούς θανάτων. Άρα κάποια άλλη εξήγηση πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να έχουμε λοιπόν μια συγκεκριμένη εικόνα των ουσιών που καταγράφονται σε κάθε συγκεκριμένο περιοχή. Δεν μπορούμε να λέμε ότι όλα τα ζυζωνιοκτώνα κάνουν κακό στην μέλισσα. Υπάγονται σε μια αυστηρή διαδικασία έγκριση στα ζυζωνιοκτώνα. Με στόχο βέβαια και την επαλήθευση ότι δεν απειλούν τη ζωή της μέλισσας η οποία είναι τόσο σημαντική για την επικονίαση, για την ευρωπαϊκή γεωργία δηλαδή. Γι' αυτό και θα πρέπει να προστατεύετε και να αντιμετωπίσετε κάθε ζημιογόνος παράγοντος. Αλλά πιστεύω ότι αρκεί η διαφοροποίηση που εισάγει η γεωργική πολιτική. Εν πάση περιπτώσει, πω σε μια καλή συνεργασία με την συγκήτρια, με τη συντάκτρια της χρωμοδότης, με τους σκιώδης συντάκτες για την καταπολέμηση του θέμα του ανταγωνισμού, την προστασία της μέλισσας και ένα καλό ρυθμιστικό πλαίσιο για την συνέχεια της Μεσολοσοκομείας υπό άριστες συνθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σας ευχαριστώ. Eh, σας ευχαριστώ κυρία Κανέτσνα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τους συναδέλφους, τους σκιώδης, έχω μερικά σχόλια. Θεωρώ ότι το προσχέδιο που έχουμε στα χέρια μας είναι καλή βάση συζήτησης. Όμως υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία τα έχουμε παραμελήσει, δεν, εμφανίζονται στην πρόταση και ίσως ορισμένα άλλα ζητήματα να υπεραπλουστεύονται. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, πρέπει να αποφύγουμε τέτοιου τύπου υπεραπλουστεύσεις οι μέλισσες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο ε, είδος και ε, τους, τις, τις επηρεάζουν πολλοί παράγοντες. Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε ότι τη σημασία που έχει η επιβίωση των μελισσών για το περιβάλλον, ε, ακόμα και για την γεωργία σε πολλές περιοχές του κόσμου, δυνατότητα των γεωργών να παράγουν ε, τρόφιμα εξαρτάται από την επικονίαση από τις μέλισσες. Στην Τσεχία δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο τέτοιο πρόβλημα, όμω γνωρίζω ότι σε άλλε χώρε έχει παρατηρηθεί σημαντική μείωση του αριθμού των μελισσών και πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Είναι και μια ο αριθμός των μελισσών ε, εξαιρετικά ευαίσθητη ένδειξη για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το φυσικό περιβάλλον. Και τα φυτοφάρμακα της βλάπτουν και το αρσενικό και άλλοι χημικοί παράγοντες που υπάρχουν στο περιβάλλον και που θα έπρεπε να μας ανησυχήσουν όταν βλέπουμε ότι πλήττουν τις μέλισσες. Τις μέλισσες δεν τις χρειαζόμαστε μονάχα για το μέλι είναι μόνο ένα από τα ε, αγροτικά προϊόντα στα οποία συνεισφέρουν οι μέλισσες, ίσως είναι το πιο γνωστό, το πιο προφανές, αλλά στην πραγματικότητα ε, συνεισφέρουν σε πάρα πολλά άλλα. Ακόμα και σε σε φαρμακευτικά προϊόντα όπως ε, η πρόπολη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ε, ένα σύστημα ελέγχου, παρακολούθησης μάλλον αυτών των ε, διαδικασιών, αυτών των εξελίξεων και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να θεσπιστεί για τον τομέα της μελισσοκομείας. Ακόμα πιο σημαντικό είναι να ελέγξουμε του ε, το εισαγόμενο μέλη από τρίτες χώρες. Πολλές φορές δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την ασφάλεια και για την ποιότητα αυτού του μελιού. Όμως αυτά τα προϊόντα κυκλοφορούν στην νέα αγορά. Άρα οφείλουμε να λάβουμε μέτρα, γιατί όσες φορές έχουν γίνει έλεγχοι, μάλλον πολλές φορές που έχουν γίνει έλεγχοι, έχουμε βρει ότι ε, το μέλι αυτό δεν τηρούσε τα πρότυπα της ε, Ένωσης. Θα προτείνουμε ορισμένες τροπολογίες ελπίζω η συζήτηση αυτή να μην πολιτικοποιηθεί, να γίνει ιδεολογική, γιατί φαντάζομαι πως όλοι θέλουμε να επιβιώσει η ανθρωπότητα και όλοι αναγνωρίζουμε ότι οι μέλησες είναι απαραίτητες για να γίνει αυτό. Ελπίζω λοιπόν και ζητώ και από τους συναδέλφους να φροντίσουμε να μην ε, περιχαρακωθούμε σε πολιτικού χαρακτήρα επιχείρηματα. Οι μελισσοκόμοι ε, στην Ευρώπη έχουν περιμένει πάρα πολύ καιρό για να αναλάβουμε τέτοιου τύπου μέτρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Εύη. Ευχαριστώ πρόεδρε να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανα και αντίθετα από τους συναδέλφους αντιλαμβάνομαι ότι η διαφορά μεταξύ μιας γνωμοδότησης και μια ε, μια έκθεση είναι μεγάλη, πολύ μικρό, ε, οπότε κατά την απόψή μου αυτό που προτείνει η εισηγήτρια με βρίσκει σύμφωνη σε μεγάλο βαθμό θα υποβάλουμε τροπολογίες ώστε να υπογραμμιστεί ο θεμελιώδης ρόλος ε, των ε, ε, μελισσών στον επικονιασμό, όχι μόνο για ολόκληρο το οικοσύστημα, αλλά και για την διατροφή μας και για την, ασφάλεια, για την τροφική ασφάλεια. Υπάρχει μια μελέτη του ΙΣΦΑΟ του 2016 που αποδεικνύει ότι η Μέλισσε βοηθούν στη βελτίωση της απόδοσης των καλλιεργιών. Ειδικότερα οι μικροί γεωργοί θα μπορούσαν να αυξήσουν την απόδοση των καλλιεργιών τους έως και 25% δωρεάν ουσιαστικά, απλά βελτιώνοντας ε, ε, τους επικονιαστές αυτούς. Αυτό φυσικά θα πρέπει να οδηγήσει σε πολλές σκέψεις περί των γεωργικών πολιτικών που ασκούμε εδώ στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Ε, άλλες που θα στείλουμε θα προσπαθήσουν να ενισχύσουν αυτό που λέει καθαρά η συγγήτρια ότι πρέπει να αναγνωριστεί ότι είναι απαραίτητο να απαγορευτούν τα νοικοτινοειδή. Ξέρουμε ότι η Ευρώπη έχει κάνει μικρά βήματα προς τα εμπρός, αλλά απομένουν πολλά να γίνουν. Ε, για να ανταποκριθούμε σε ανησυχίες ε, χιλιάδων πολιτών μάλιστα, μέσω πολλών καταγγελιών και αναφορών ε, προς τα ευρωπαϊκά όργανα. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να κάνουμε αυτό το βήμα προ τα εμπρό, γιατί ξέρετε δεν υπάρχουν πια αιτιολογίε. Είναι εκατοντάδε πλέον οι μελέτε που το αποδεικνύουν ότι το ποσοστό θνησιμότητας των μελισσών που εκτίθενται ε, σε αυτά τα ε, νοικοτινοειδή είναι 30% ε, μεγαλύτερο από τις μη εκτεθειμένες, με τους μη εκτεθειμένους πληθυσμούς. Οπότε πρέπει να κάνουμε κάτι σε αυτό το μέτωπο. Για να κλείσω, να πω ότι ο τομέας της μελισσοκομείας πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της οικολογικής και γεωργικής μετάβασης που συντελείται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να βασίσουμε τη γεωργία μας σε φυσικές δυνάμεις και σε βιώσιμες πρακτικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, χρόνια τώρα, για να μην πω δεκαετίες, ε, εκφράζει τις ανησυχίες της για τα ζητήματα αυτά του μελισσοκομικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ομάδα μου, οι πιο παλιοί εδώ στο Κοινοβούλιο θα θυμούνται την πρώην συνάδελφο Άστριντ Λούλινγκ, η οποία ε, φό εκφωνούσε πύρινους λόγους πάντοτε στα θέματα αυτά. Τώρα λοιπόν πια έχει έρθει η ώρα η Γεωργία να υπολογίσει τα σοβαρά τον το με αυτόν και τις προκλήσεις που φέρνει μαζί, που, που συνεπάγεται. Για το θάνατο των μελισσών δεν θα επεκταθώ. Τα κάλυψαν οι συνάδελφοι και έχουμε συστήσει πολλές φορές και στην Επιτροπή μας. Η παραγωγή ε, μελιού ως εκ τούτου στην Ευρώπη είναι ελληματική, αναγκαζόμαστε να εισάγουμε. Ξέρουμε ότι η παραγωγή των τρίτων κρατών αυτή τη στιγμή δεν τηρούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία και αυτό το οποίο παίρνει το χαρακτηρισμό μέλη εισαγωγής δεν είναι μέλη. Καθήκον μας είναι να προστατεύσουμε τον καταναλωτή και δει με πολύ συγκεκριμένο και αυτό τρόπο. Υποστηρίζω λοιπόν αμέριστα τις ε, παρατηρήσεις των της σκιώδους εισηγήτριας της ομάδας μου, της κυρίας Μαγκίνες. Είναι σημαντικό πιστεύω να διευκρινιστούν κάποια θέματα Περισσότερο όμως ακόμη να υποστηρίξουμε το μέλι και την εικόνα του. Πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίε στη Γαλλία, ήδη και στη Νότια Γαλλία υπάρχουν πρωτοβουλίε εξαιρετικέ εδώ και χρόνια και μοναδικές. Ε, πρέπει να πάρει πιο επαγγελματικό χαρακτήρα το επάγγελμα του μελισσουργού, ε, να διευκολυνθεί η γενετική επιλογή με βάση την κατάλληλη κατάρτιση και γνώσεις. Βλέπετε ότι υπάρχει μια σειρά από επιχειρήσεις που μπορούμε να υποστηρίξουμε σε διάφορους ε, άξονες και έχουμε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκροστέτ. Κυρία Ρης. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα θυμίσω και εγώ πως και η κυρία Γκροστέτ την Αστρίτ Λιούλινγκ που ξέρετε πολύ με με τρυφερότα αποκαλούσαμε εδώ μέσα Μάγια η Μέλισσα. Ε, όντως δεν είναι πολύ καιρό που ήταν ακόμα εδώ. Η κυρία Γκροστέτ ε, είναι μεταξύ εκείνων που συνέπραξαν στην διοργάνωση της Big Week, ε, της εβδομάδας της Μέλισσας ε, πριν το καλοκαίρι, με συμμετοχή εκπροσώπων των μελισσουργών και μελισσοκόμων και υποστήριξη προς μια ιδέα για μια γνώμοδότηση που βέβαια ξέρουμε ότι χρειάζεται κάποια συμπλήρωση, λείπουν κάποια σημεία. Ως προς την ουσία θα έλεγα ότι είναι καλό, όπως είπε και η κυρία Μαγκίνες, να συνενώσουμε λίγο τα ε, σημεία της πρότασης ώστε να μην έχουμε επαναλήψεις πολλές, το 5 και το 10 παραδείγμα, το 2 και το 5 παραδείγματα. Ε, κάποια άλλα σημεία που ε, είναι πολύ σημαντικά, ε, όπως σε παραδείγματι τα νεονικοτινοειδή. Μπορεί να τα είπε στην ομιλία της η συντάκτρια, αλλά δεν τα έχει στο κείμενο. Και πρέπει να μπουν, γιατί δεν είναι κάτι το αμεληταίο. Είναι πολύ τοξική ουσία για τις μέλισσες. Και έχει καταχωριστεί ως τέτοια από το 2013. Υπάρχει και ένα τεράστιο ε, μια τεράστια αναφορά με χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες υπογραφές από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκφράζουν με τον τρόπο αυτό την ασυχία τους. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να μελήσουμε και πάντως όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάποια άλλα σημεία που δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τα καλύψουμε με τις τροπολογίες, κλιματική αλλαγή, καταστροφή ενδιαιτήματος, μια σειρά από ε, επιζωοτίες όπως η βαρόαση, νομίζω ότι θα πρέπει να καλυφθούν. Ε, επίσης, δεδομένα και έρευνα, η Επιτροπή και από τελευταία, τον τελευταίο κατάλογο των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών σας, καταγράφει χίλιες από τα 2.000 από τα 2.000 είδη μέλισσας ως ε, απειλούμενα με εξαφάνιση. Επομένως, βλέπουμε ότι είναι η κατάσταση πάρα πολύ σοβαρή. Χρειαζόμαστε στατιστικά επακριβή, καλής ποιότητας, για να έχουμε μια συγκεκριμένη εικόνα του κινδύνου. Αυτό άλλωστε ζητά και η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα που ξεκίνησε με την εβδομάδα της Μέλισσας ε, ε, τον Ιούνιο. Αυτές ήταν οι πρωταρχικές μου παρατηρήσεις. Πάνω σε αυτές θα στηρίξω τις τροπολογίες μου και προσβλέπω σε συνεργασία με όλες ε, εκείνες, γυναίκες βλέπω, ε, τις συναδέλφους ε, που οργάνωσαν την ε, εβδομάδα της Μέλισσας. Δεν ξέρω γιατί ήταν μόνο γυναίκες, θα σκοπούμε σκόπιμο να κοιτάξουμε και λίγο τι κρύβεται πίσω από αυτό. Συνεχίζουμε πάντως τη δουλειά της Άστριντ Λούλιν και ευχαριστώ. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Σάπς, πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω επίσης και τον εισηγητή που υποβάλλει αυτές τις σημαντικές για τον τομέα της μελισσοκομείας συστάσεις που βρίσκονται και στην καρδιά των ανησυχιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γνωρίζουμε ότι οι μέλησες είναι ευαίσθητες. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να τις φροντίσουμε γιατί είναι απαραίτητες για τον επικονία, την επικονίαση για την αναπαραγωγή των φυτών και για τη γεωργία, καθώς επίσης και για την παραγωγή ε, μελισσοκομικών προϊόντων, μελιού και λοιπόν. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η μελισσοκομεία είναι σημαντικός τομέας της περιφερειακής αγροτικής οικονομίας σε διάφορες περιοχές των κρατών μελών. Θα θέλαμε λοιπόν να υποστηρίξουμε τα φυσικά οικοσυστήματα των μελισσών, αυτών των σημαντικών φυσικών επικονιαστών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου υπάρχουν προβλήματα με την ε, επάρκεια των τροφίμων. Θα ήθελα να προσθέσω κάποια στοιχεία στον προβληματισμό σας. Η κυρία Μακίνες ήδη ανέφερε τι διεμήφθη στην Επιτροπή Κομμάτρη. Θα ήθελα να επισημάνω ότι μέσω της κοινή αγροτικής πολιτικής υποστηρίζουμε σημαντικά τους μελισσοκόμους. Υπάρχουν κονδύλια που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό για την ε, υποστήριξη προγραμμάτων μελισσοκομείας της τάξης των 36 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι αυτό έχει αυξήσει τα μελίσια σε ορισμένες ορατικές περιοχές, έχει τόση αποτελέσματα, έχει ενθαρρύνει τον τομέα της μελισσοκομείας και στην πράξη. Ε, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε λοιπόν ότι η κοινή αγροτική πολιτική προβλέπει τρία διαφορετικά χρηματοδοτικά μέσα για την προστασία του περιβάλλοντος. Η κυρία Μακίνες αναφέρθηκε στις λεγόμενες ενέργειες για το πρασίνισμα, το greening. Ε, υπάρχουν όμως και στοιχεία στην, ε, στον έλεγχο που γίνεται για τη διασταυρωμένη συμμόρφωση. Η προστασία του περιβάλλοντος επίσης προβλέπεται και στα διορθωτικά ταμεία και στα περιφερειακά ταμεία. Είναι κριτήρια ε, που ε, προβλέπονται και συμπεριλαμβάνουν ε, και την προστασία των μελισσών. Βέβαια, συμφωνώ μαζί σα ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το προσέξουμε ακόμα περισσότερο, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ζυζανιοκτώνα και τα φυτοπροστατευτικά μέσα. Η διαδικασία για τις εγκρίσεις αυτών των προϊόντων είναι εξαιρετικά αυστηρή γνωρίζετε ότι δίνεται έγκριση σε ένα ε, προϊόν μόνο εάν αποδειχθεί ότι το προϊόν δεν εγκυμονεί κινδύνους ε, ούτε για τους ανθρώπους ούτε για τα ζώα. Παρατηρούμε λοιπόν την εξέλιξη της κατάστασης ε, αυτές τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων παραγόντων του, περιβαλλοντικών και της αναπαραγωγής των μελισσών και α, αντιστοίχως προσαρμοζόμαστε. Αναφερθήκατε στα νεονικοτοειδή. Ε, είναι ένα χημικός παράγοντας στον οποίο, από, για τον οποίο ζητήσαμε γνώμοδότηση από την ΕΦΣΑ έτσι ώστε να ακολουθήσουμε μια ε, επιστημονική προσέγγιση, να μην ε, πάμε ούτε προς τη μία ούτε προς την άλλη κατεύθυνση ε, χωρίς επιστημονικά δεδομένα στα χέρια μας. Όσον αφορά τώρα τον έλεγχο για την ποιότητα του μελιού, οποιαδήποτε είδος μελιού τίθεται στην ευρωπαϊκή, στην στήν αγορά, έχει ελεγχθεί, υπάρχει πρόβλημα ορισμένες, σε ορισμένες περιπτώσεις για τα, τη μέτρηση των σακχάρων. Ναι. Και προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τους ειδικούς στον κλάδο αυτό για το ζήτημα. Έτσι ώστε να καταρτιστεί για το 2015, 2017 μάλλον καταρτίστηκε το 2015-2017 ένα νέο πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την, για την έλεγχο αυτών και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις τρίτες χώρες είναι ευρύτατα διαδεδομένη η πρακτική να προστίθεται ζάχαρη στο μέλι που τίθεται στην αγορά. Συνεργαζόμαστε εδώ με τις αρχές των κρατών μελών, γιατί εκείνες είναι που κάνουν τους ελέγχους. είναι οι εθνικές αρχές για την ασφάλεια των τροφίμων που εξασφαλίζουν την ποιότητα του μελιού, μεταξύ άλλων. Και πάλι λοιπόν ε, θα κάνω μια έκκληση σε όλους τους εμπλεκόμενους, σε όλους τους ενδιαφερόμενους να συνεργαστούν, γιατί μόνο έτσι θα τα καταφέρουμε. Να δώσουμε μια λύση που θα γίνει αποδεκτή από τους πολίτες στην Ευρώπη και ταυτόχρονα από τους ε, δραστηριοποιούμενους στον κλάδο και τους μελισσοκόμους. Ευχαριστώ. Κύριε Ντονάνο, εισηγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θα απαντήσω, βέβαια, σε κάθε παρέμβαση για την κυρία Μακίνες. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις της. Σας βεβαίως μπορεί να τροποποιηθεί ενδεχομένω η δομή για την ΚΑΠ ασφαλώς θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προστατευόμενες περιοχές, αλλά και άλλες, καθώς και τα ε, αντίξω αποτελέσματα που μπορεί να προξενηθούν ε, από την ΠΑΚ, ε, ΚΑΠ και βεβαίως και οι άγρες ε, μέλησες. Για τον συνάδελφο χρειαζόμαστε περισσότερα μέσα. Θα σημειώσετε ότι δεν μιλώ μόνο για ζυζανιοκτώνα ε, για τις μέλισσες και ενώ η γλυφοζάτη ακόμη χρησιμοποιείται παρότι ε, είναι επικίνδυνη συγκεκριμένα για τις ε, μέλισσες, για την κυρία Κονεσλέν θέλω να υιοθετηθεί η έκθεση μου για το καλό της μέλισσας και άρα για, το μέλλον της ανθρωπότητας και γι' αυτό προτείνω μια συνετική βάση εργασίας. Μιλώ για το ως προϊόν, οτιδήποτε είναι γύρω από την ε, κυψέλη. Ε, και βέβαια τα προϊόντα μπορεί να προκύψουν από το μέλι, πρόπολη κτλ. Εάν γίνει η πολιτική αντιπάθεση γύρω από αυτό δεν θα οφείλεται σε δική μου πρόθεση. Για την άλλη συνάδελφο, ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις της και περιμένω τις τροπολογίες για να βελτιωθεί η έκθεσή μου. Έτσι άλλωστε εννοώ εγώ την δουλειά και τη συνεργασία με τους συναδέλφους. Με τους πολίτες επίσης περιμένω τις ερωτήσεις τους, γιατί με τις ερωτήσεις που απευθύνουν στους ευρωβουλευτές βελτιώνονται οι προτάσεις. Ε, κυρία Γκροστέτ, όπως βλέπουμε, με ρημνά ιδιαίτερα για τις μέλισσες, γιατί όχι, αλλά μην ξεχνάμε και ότι η ΚΑΠ με την υπερβολική απέτηση για παραγωγή δεν μπορεί να επιτρέψει στις την επιβίωση της μέλισσας. Η λιφοζάτη, όπως και άλλα συζανιοκτώνα ε, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο συμβατό με τη διαφύλαξη του είδους. Για την κυρία Ευχαριστώ να αναφερθούν τα νέα νοικοτινοειδή, εκ των οποίων όμως μέρος ε, αυτή τη στιγμή είναι απαγορευμένη η ουσία. Ε, στόχος μου είναι, όπως καταλαβαίνετε, να ε, προκύψει μέσα από συμφωνία με τις ομάδες η έκθεσή μου. Βεβαίως εγώ θα αναφέρω τη Βαροάση και άλλα και άλλες επιζωτίες που απειλούν τη μέλη, όπως και τα νοικοτινοειδή στις τροπολογίες μου, κομισιόν. Η η υπερβολική ε, παραγωγή, η εντατικοποίηση της παραγωγής που ε, προκύπτει από την ΚΑΠΑ είναι ο κύριος κίνδυνος για την μέλισσα. Τα λίγα, λίγες εκατοντάδες χιλιάδες που μπορεί να δώσετε για τη μέλισσα είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στα εκατομμύρια ευρώ που διαθέτουν τα μεγάλα κράτη, κυρίως όπως η Γαλλία στον ευρωπαϊκό προπολογισμό και χρειάζεται μια ουσιαστική προσέγγιση. Η μέλισσα που έχει κάποια ψήγματα επιδοτήσεων. Σας ευχαριστώ. Τροπολογίες 3 Οκτωβρίου. 11 η ώρα. 19 Οκτωβρίου, Επιτροπή Ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ θερμά και καλό σας μεσημέρι. Next meeting, 11th Okay?